Αγαπητοί συνάδελφοι, με συγχωρείτε, επειδή υπήρξε μία ασθένεια. Δεν είχε να κάνει με την... Ε, η καθυστέρησή μου λοιπόν οφείλεται σε αυτό, δεν είχε να κάνει με την ε, γιορτή της μπύρας. Λοιπόν, ανακοινώσεις της Προέδρου. Λοιπόν, έχουμε μετάφραση, έχουμε μετάδοση στο ίντερνετ, δεν έχω τίποτα να σας πω. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 της μέρης διάταξης, ετήσια έκθεση 2018 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ε, χαίρομαι που έχουμε σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την 30η ετήσια έκθεση για την προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση αυτή. Θέλω να συνδέσω αυτή την ετήσια έκθεση με το ευρύτερο πλαίσιο των ε, μέτρων εκείνων που λάβαμε τα τελευταία χρόνια υπό την ευθύνη μου με σκοπό την ε, καλύτερη προστασία των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ως Κομισιόν, σε συμφωνία και μαζί σας, τα τελευταία χρόνια υποβάλαμε σημαντικές ε, προτάσεις σε όλους τομείς του ευρωπαϊκού προπολογισμού και για τα έσοδα και για τις δαπάνες. Και η έγκριση των μέτρων αυτών από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο άλλαξε σημαντικά το τοπίο της ε, καταπολέμησης της απάτης. Στην ομοθεσία εγκρίθηκαν δύο σημαντικές ε, πρωτοβουλίες που ενίσχυσαν την ε, προστασία των οικονομικών συμφερόντων από την σκοπιά του ποινικού δικαίου. Πρώτον ήταν η οδηγία για την ποινική δίωξη των περιπτώσεων απάτης ε, ει βάρο των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση, η οδηγία PIF, καθώς και ο κανονισμός για την ενισχυμένη συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Με την ε, δημιουργία, την ίδρυση τη Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, εσείς άλλωστε πριν από λίγες μέρες ψηφίσατε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άλλαξε θεμελιωδώς πλέον το νομικό πλαίσιο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Συγκυλία είναι ένα θεσμικό όργανο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί αυτεπάγγελτα να ξεκινά δικαστικές έρευνες καθώς και να απευθύνεται να προσφεύγει στα εθνικά δικαστήρια για εικαζόμενες ε, παρατυπίες ή αδικήματα. Αυτή τη στιγμή στο μηχανισμό αυτό συνεργασία συμμετέχουν 22 από τα 28 κράτη-μέλη, ενώ και άλλα ε, κράτη-μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στην μορφή αυτή της συνεργασίας. Εγώ και η συνάδελφή μου, η κυρία Γιούροβα, λαμβάνουμε διαρκώς μέτρα και κατευθυνόμαστε προς το να πείσουμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ακριβώς για να ολοκληρωθεί αυτή η μορφή συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν αποτελεί ένα νέο φορέα ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο της καταπολέμησης απάτης. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι έπρεπε να προσαρμοστεί και το modus operandi του Όλαφ. Πρέπει βεβαίως να υπάρξει μια διάκριση των αρμοδιοτήτων, αλλά και να διαμορφωθεί ε, και να ρυθμιστεί νομικά η συνεργασία μεταξύ του Όλαφ και της Ευρωπαϊκής ε, Εισαγγελίας. Νομίζω ότι ακριβώς χάρη στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεχίσουμε να χρειαζόμαστε αυτό το ανεξάρτητο όργανο, τον Όλαφ, που στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα μπορεί να επιτελεί τα δικά του καθήκοντα. Και για να καταστήσουμε την προστασία από την απάτη ακόμη πιο αποτελεσματική, εγώ ήθελα να παράσχω στον Όλαφ εκείνα τα εργαλεία ώστε να μπορεί η υπηρεσία αυτή να αντιμετωπίζει όλο και πιο σύνθετες μορφές της απάτης. Πέρσι υποβάλαμε και μια πρόταση τροποποίησης της νομικής βάσης του Όλαφ, η οποία διαβιβάστηκε βεβαίως και σε εσά και στο Συμβούλιο ώστε να λαμβάνεται πλέον υπόψη η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προκειμένου να καταρτιστεί αποτελεσματικότερο το έργο του Όλαφ καθώς και να ε, ρυθμιστεί για το μέλλον με σαφέστερο τρόπο η διάκριση των αρμοδιοτήτων. Έκθεση PIF 2018 καταδεικνύει την πρόοδο που ε, την ε, τελευταία χρονιά στον τομέα της καταπολέμησης ε, της απάτης και των παρατυπιών, καταδεικνύει όμως και τους τομείς στους οποίους χρειάζεται βελτίωση. Ωστόσο, για την προστασία της, ε, του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν είναι αρμόδια μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καθώς περίπου το 75% των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων υπόκειται σε διαχείριση σε επίπεδο κράτους μέλους, είναι εύλογο αυτό. Αυτή η κοινή ευθύνη λοιπόν εκφράζεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη αλλά και με τις περιφέρειες και τις ε, τοπικές κοινότητες υποβάλλει μια έκθεση για την προστασία των μέτρων που έχουν ληφθεί για την, προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Σε αυτή την έκθεση που υποβάλλεται εδώ και 30 χρόνια, η Κομισιόν συντάσσει συστάσεις προς τα κράτη-μέλη για το τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για να αρθούν προβλήματα τα οποία έχουν ε, εντοπιστεί. Φέτος λοιπόν, με αφορμή την 30η ε, επέτειο της υποβολής αυτής της έκθεσης, κάνουμε και μια ανασκόπηση στην ε, έκθεση που σας υποβάλλουμε. Και εκεί καταδεικνύεται και η πρόοδος που έχει γίνει στη διάρκεια των δεκαετιών και ιδίως την τελευταία ε, πενταετία. Καταφέραμε πολλά. ο εντοπισμός το 2018 ε, των παρατυπιών αυξήθηκε κατά 15%. Ενώ οι μη εντοπιστήσεις ε, παρατυπίες ε, μειώθηκαν ε, κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζουμε ότι αυτή η θετική τάση αποτελεί άμεση επίπτωση, συνέπεια της υλοποίησης των προταθών, ε, με, ε, ε, των μέτρων από την Κομισιόν για την καταπολέμηση της απάτης. Βεβαίω, ξέρουμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά ακόμη. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι η προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι εξαιρετικά σημαντικός, ιδίω σε μια εποχή στην οποία έχει τεθεί σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη των πολιτών μας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η προστασία των οικονομικών συμφορώντων περιλαμβάνει ολόκληρο τον ε, κύκλο της καταπολέμησης απάτης. Από την πρόληψη έως ε, την αποκάλυψη, την ε, έρευνα, την ποινική δίωξη, έως και την ανάκτηση και την επιβολή κυρώσεων. Και με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή τη διαδικασία μάλλον, περιλαμβάνονται διάφοροι φορείς στο πλαίσιο της, ε, του σχεδιασμού των ε, προγραμμάτων, της σύλληψη των προγραμμάτων, τους ελέγχους και τις έρευνες και την ποινική οδίευση. Δυστυχώς όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά και εντός του ίδιου κράτους μέλους πολλές φορές ε, δεν είναι τα πράγματα πάντοτε ομοιόμορφα για το πώς αντιμετωπίζεται η απάτη βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, ποιο είναι το επίπεδο και το εύρος συνεργασίας με τον Όλαφ ή σε ποιο βαθμό ακολουθούνται οι συστάσεις του Όλαφ. Και εδώ προσπαθούμε πάντοτε να ερχόμαστε σε διαβούλευση, να ασκούμε πίεση, γιατί δεν είναι σωστό ε, στην ε, χρήση, η χρήση των ε, κονδυλίων να παρουσιάζει τέτοιες μεγάλες διαφορές, όπως βεβαίως και η καταπολέμηση της κατάχρησης αυτών των κονδυλίων. Πρέπει να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και γι' αυτόν το λόγο και στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2021 θα εντάξουμε διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης και ελπίζουμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σύντομα εντός του 2019 ή έως το 2020 να εγκρίνουν την ε, προαναφερθήσα τροποποίηση του κανονισμού για τον Όλαφ. Αυτή η προτινόμενη τροποποίηση του κανονισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια στενή συνεργασία μεταξύ του Όλαφ και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Και αυτό είναι μια αναγκαία συνθήκη για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία αλλά και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του ευρωπαϊκού συστήματος καταπολέμησης απάτης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει αποτελεσματικότερη ποινική δίωξη των περιπτώσεων αναπάτης στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των εθνικών τους διαδικασιών. Όμως, για να έχουμε ολοκληρωμένη προστασία του προπολογισμού, δεν έρχονται μόνο ποινικά, χρειάζονται και διοικητικά μέτρα. Και γι' αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Όλαφ έχουν διαφορετικές μεν αλληλοσυμπληρώμενες όμως υποχρεώσεις και καθήκοντα. τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατόπιν σύστασης ε, του Όλαφ μπορούν ε, να προβαίνουν σε άμεση ανάκτηση ποσών τα οποία έχουν ε, υπάρξει αντικείμενο κατάχρησης χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν σύνθετες και συχνά χρονοβόρες ποινικέ διαδικασίες έως ότου ολοκληρωθούν αυτές. Όπως είπα, σας ε, απευθύνω έκκληση σύντομα να εγκρίνετε αυτή την τροποποίηση του κανονισμού για τον Όλαφ και έτσι να αντικατοπτριστεί και η βασική συλλογιστική της Κομισιόν. Δηλαδή να έχουμε έναν ισχυρό Όλαφ, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι σε θέση να επιτελεί τα καθήκοντά του, και που θα μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Ξέρω ότι οι επικείμενοι τριμερείς διάλογοι δεν θα είναι εύκολοι, διότι μεταξύ άλλων και οι εντολές διαπραγμάτευσης ε, των, ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι αρκετά διαφορετικές. Όμως ο στόχος μας είναι ίδιος. Θέλουμε να ε, προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για το λόγο αυτό η Κομισιόν και η νέα Κομισιόν θα υποστηρίξει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση, να εξευρεθεί ένα συμβιβασμός και να μην σπαταληθεί χρόνος, γιατί θέλουμε από του χρόνου και όλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλάβει τα καθήκοντά της και θα πρέπει να υπάρχει ε, και ένας, ε, ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα ανταποκρίνεται και στα μελλοντικά καθήκοντα. Η νέα στρατηγική της Κομισιόν για την καταπολέμηση της απάτης CAFS, Commission Anti-Fraud Strategy. Αυτός ο τρίτος πυλώνας ε, των εργασιών μας εξασφαλίζει ότι μπορούμε να παρακολουθούμε ε, τις ε, διαρκώς μεταβαλλόμενες μορφές της απάτης. Οι απαταιώνες προσαρμόζονται διαρκώς και χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να επιτύχουν τους στόχους τους. Και αυτός είναι ο λόγος που τον Απρίλιο του 2019 η Κομισιόν παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την καπτολέμηση απάτη. Έχει δύο άξονε: Εμβάθυνση των γνώσεων τη Κομισιόν όσον αφορά του κινδύνου απάτη και ενίσχυση τη υπηρεσιακή ε, εποπτείας εντό τη Κομισιόν. Και εδώ η δική σα επιτροπή έχει πολλές φορές ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τις αιτίε ε, των περιπτώσεων απάτης ε, εις βάρος Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, καθώς και για τις διαφαινόμενε τάσεις. Και το χαιρετίζω αυτό. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις αναλυτικές ικανότητες του Όλαφ και να δώσουμε στην υπηρεσία αυτή τον χαρακτήρα ενός κέντρου γνώσεων για την καταπολέμηση απάτης. Γιατί ένα τέτοιο κέντρο γνώσεων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης και να υποστηρίξει έγκαιρα και αποτελεσματικά τόσο τις υπηρεσίες της Κομισιόν όσο και τα κράτη-μέλη με στήριξη και με συμβουλές. Και για να ε, υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή την κατεύθυνση, θεσπίσαμε και την ε, ενδοϊπηρεσιακή εποπτεία εντός της Κομισιόν. Η νέα στρατηγική ενισχύει δηλαδή τον ρόλο του Όλαφ στον ε, συντονισμό των μέτρων καταπολέμησης απάτης μεταξύ των μεμονωμένων υπηρεσιών της Κομισιόν. Εδώ και τέσσερα χρόνια η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν εθνικές ε, στρατηγικές για την καταπολέμηση τη απάτη, για να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι σήμερα, μόλις 11 κράτη-μέλη έχουν καταρτήσει τέτοιες εθνικές ε, ε, στρατηγικέ και τι έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν. Αλλά τρία κράτη-μέλη έχουν τέτοιες εθνικές στρατηγίες, δεν τις έχουν κοινοποιήσει. Τέσσερα ακόμη ε, βρίσκονται στο στάδιο της κατάρτισης μια τέτοια μιας τέτοιας στρατηγικής. 18 κράτη-μέλη λοιπόν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα έχουν τέτοιες στρατηγικές και θα τις έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν. Στην έκθεση PIF ε, τονίζουμε για άλλη μια φορά την σύστασή μα προ τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν τέτοιε εθνικέ στρατηγικέ για την καπιτολέμηση τη απάτη. Και η δική σας Επιτροπή έχει, κάνει, έχει απευθύνει σχετική έκκληση στα κράτη-μέλη και βεβαίως αντίστοιχες εκκλήσεις έχει κάνει και ε, το ελεγκτικό συνέδριο στην ειδική έκθεση με τίτλο «Καταπολέμηση της απάτης στις δαπάνες συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Θεωρώ λοιπόν ότι η κατάρτιση εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης απάτης ε, είναι ένα σημαντικό βήμα στις κοινέ μας προσπάθειες για την καταπολέμηση της απάτης και των παρατυπιών σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Ευρωβουλευτέ, στην διάρκεια της θητείας μου ως αρμόδιος για τον Όλαφ, δημιουργήσαμε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την βελτίωση της ε, καταπολέμησης απάτης και από τα κράτη-μέλη, ε, από τα οποία λάβαμε υποστήριξη και από τα κράτη-μέλη τα οποία λαμβάνουν μεγάλα ποσά του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Η σημαντικότερη προϋπόθεση ε, βεβαίως Βεβαίω για την επιτυχία αυτή τη στρατηγική, αυτού του νομικού πλαισίου που δημιούργησε η Κομισιόν, είναι η πρόβλεψη αναγκαίων πόρων. Είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι πόροι, αν διατεθούν, θα πιάσουν τόπο γιατί πολλά από τα χρήματα τα οποία ε, γίνονται αντικείμενο κατάχρησης θα επανέλθουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αφενός αυτό, αφετέρου δε θα μας βοηθήσει μια τέτοια επένδυση γιατί θα αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Η έκθεση PIF του 2018 δείχνει ότι οι προσπάθειές μας στέφτηκαν από επιτυχία, με επιτυχία. Και σε αυτό μπορεί να, να βασιστεί και η νέα Κομισιόν. Ευχαριστώ εσάς και την κυρία Γκρέσλε, την πρώην πρόεδρο της Επιτροπής, για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξη. Θεωρώ ότι και η κριτική που μας ασκήσατε ήταν πάντοτε πολύ γόνιμη και επικοδομητική και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για την συζήτηση που θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Γκρούση να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ότιγκερ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκθεσή που μας παρουσιάσατε. Για μένα είναι όλα αυτά πολύ καινούρια και είναι μεγάλη τιμή που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, να ασχοληθώ με αυτόν τον κόσμο. Διάβασα όλες τις εκθέσεις μέχρι και πριν από 30 χρόνια και, και μετά λέει ότι η καταπολέμηση της ε, απάτης είναι βασισμένη στην ανάγκη για συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς αυτή τη συνεργασία η καταπολέμηση της απάτης ε, θα αποτύχει. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα είναι προϋπόθεση. Ούτως ώστε η καταπολέμηση της απάτης να επιτύχει. Αυτό όμως ε, λείπει στην έκθεσή σας. Αναφέρονται πολλά πράγματα. Όπως λέει και το ε, άρθρο τη συνθήκη για, για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενημερώνεται για το τι έχετε κάνει κάθε χρόνο κατά τη απάτη. Πολλά πράγματα. Πράγματα μου έκανα τεράστια εντύπωση. Θα προτιμούσα βέβαια να τα έχω διαβάσει στα γερμανικά. Τα καταλαβαίνω καλύτερα από τα αγγλικά, αλλά τέλο πάντων. Ε, τα κατάφερα και το πάλεψα. Είδα πολλά προγράμματα που θέλετε να εισαγάγετε. Το τελευταίο το έντις. Στο τέλος λέτε αυτό το σύστημα για την έγκαιρη ανείχνευση και αποκλεισμό. Είναι ένα σύστημα λοιπόν έγκαιρης προειδοποίησης. Πού βασίζεται. Στα άρθρα 135-145 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και αν κοιτάξει τα άρθρα αυτά κανείς διαπιστώνει ότι δημιουργείται μια τεράστια δομή, πολύ περίπλοκη κανονιστική διαδικασία και βλέπω στην έκθεσή σας ότι πέρυσι ότι εντοπίσατε έξι περιπτώσεις μέσω αυτής της υπηρεσίας. Έξι περιπτώσεις. Και το 2017 δύο περιπτώσεις και φέτος λέτε ότι εντοπίσατε 8 περιπτώσεις. Υπάρχει μια ανισορροπία. Δηλαδή γίνεται τέτοια τεράστια δαπάνη, δημιουργείται ένα ολόκληρο όργανο με υπαλλήλου υψηλού επίπεδου και τι κάνουν, ασχολούνται με έξι περιπτώσεις. Όντως ισχύουν αυτά τα νούμερα. Μία ερώτηση. Ε, δυσαναλογία λοιπόν και τη βλέπω και σε άλλα σημεία. Λέτε ότι επιδιώκεται με ηλεκτρονικό τρόπο, με διάφορες μεθόδους εντοπισμού, με διάφορες βαριές διαδικασίες. Προσπαθείτε να εντοπίσετε απάτες. Αλλά, όπως είπατε, χρειάζεται συνεργασία. Αλλά δεν βλέπω να λέτε πολλά για συνεργασία, παραλαμβάνω. Γι' αυτό θέλω να κάνω τις ερωτήσεις αυτές και να μας πείτε κατά πόσο αντιστοιχούν ε, οι δομές αυτές στη διαδικασία τα οποία μέτρα λέτε ότι πρέπει να είναι και αποτρεπτικά. Δεν καταλαβαίνω τώρα εάν πραγματικά λειτουργούν αποτρεπτικά. Κάτι γενικότερο. Κάτι άλλο που δεν το είδα στην έκθεση. Οι περιπτώσεις που περιγράψατε αφορούν διάφορες ε, χώρες. Δεν βλέπω μια γενικότερη προσέγγιση που να λέει ε, πού ακριβώς προέκυψαν τα προβλήματα. Εδώ σε υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε κάποιες χώρες, σε κάποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα ήθελα μια κάποια κατανομή. Επίσης, μας εξηγήσατε ότι βελτιώθηκε πολύ κατάσταση τα τελευταία 30 χρόνια, αξιέπαινο αυτό. Αλλά, εάν τα συστήματα που έχουμε τώρα λειτουργούν σχετικά καλά και μειώθηκαν οι δαπάνες, γιατί χρειαζόμαστε τον ε, Ευρωπαίο Αγγελέα Καταλαβαίνω ότι η ερώτησή μου είναι κάπως προκλητική. Επίσης, είπατε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι τα κατάλληλα και ανάλογα. για να καταπολεμηθεί η απάτη. Όμως, σε αυτόν τον ε, ηλεκτρονικό κόσμο προσπαθούμε, προσπαθούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Η πρόεδρος. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μιλάτε ήδη 6 λεπτά. Σας παρακαλώ, έχετε μιλήσει περίπου όσο και ο Επίτροπος. Συνήθως οι εισηγητές έχουν 4 λεπτά. Και σας έδωσα και 2 λεπτά παραπάνω. Παρακαλώ τελειώνετε. Ναι, μα ρώτησα. Πόσο μπορώ να μιλήσω και μου είπαν ότι μπορώ να μιλήσω όσο περίπου και ο επίτροπο. Ίσως έγινε κάποιο λάθο. Εντάξει, θα τελειώνω. Θα τελειώνω ένα-δύο θέματα ακόμη. Γιατί έχω πάρα πολλά θέματα. Οπότε, τέλο πάντων, θα θέσω μόνο ένα ερώτημα επιπλέον. Διαφάνεια. Πολύ σημαντική για τέτοιε διαδικασίε. Πώς τα καταφέρετε να γίνονται σεβαστές οι ρήτρε του κανονισμού προστασίας ε, δεδομένων. Από τη μία πρέπει να προστατεύουμε την ε, ιδιωτική σφαίρα, από την άλλη βέβαια πρέπει να συλλέξουμε στοιχεία που είναι και προσωπικά πολλές φορές. Πώς ε, συνδυάζονται αυτά τα δύο. Κάτι ακόμη. Αναφέρεται διάφορα στοιχεία. έχουν και στοιχεία από συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα, απάτες για επιδοτήσεις. Τα στοιχεία αυτά τα συμπεριλαμβάνετε όλα στους υπολογισμού σας. Και ένα τελευταίο. Ποιος είναι ο ορισμός της απάτης, εάν μια παρατυπία είναι απάτη ή όχι. Κάνετε μεγάλες ε, διαφοροποίησεις στατιστικές. Πώς καθορίζεται, με τι κριτήρια και σε ποια φάση αποφασίζεται αν κάτι πρέπει να αποσταλεί ε, προς δικαστική δίωξη. Ε, αυτά τα λίγα. Μπορώ να σας στείλω και άλλες ερωτήσεις γραπτός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, κύριε Επίτροπε, που μας παρουσιάσατε τα θέματα αυτά και αυτό που με ικανοποίησε ιδιαίτερα είναι ότι θέλετε να δημιουργήσετε δυνατότητα πρόσβασης στην Επιτροπή, στην Όλαφ, στο ελεκτικό συνέδριο, στον Ισαγγελέα. Τι σημαίνει αυτό. Θα υπάρχει δυνατότητα κανείς ε, Έχει κανεί πρόσβαση και χωρί ε, πολλέ ε, αδειοδοτικέ διαδικασίε, γιατί αλλιώ τι έννοια έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσετε εδώ να κάνω αυτέ τι ερωτήσει. Ε, σχεδόν 10 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Αν συμφωνείτε, να απαντήσει ο Επίτροπος ε, Ίσως όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, που έκανε ο εισηγητής και μετά να πάρουν το λόγο οι επόμενοι τρεις ε, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Καταρχάς για το ερώτημα για το πώς ε, δημοσιεύεται η έκθεση. Πώς αυτή τη στιγμή η έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη σε τρεις γλώσσες και στα γερμανικά. Και με βάση τις δυνατότητες ε, των ε, μεταφραστικών μας υπηρεσιών θα μεταφραστεί τις επόμενες μέρες και στις υπόλοιπες ε, επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Είναι υποχρέωσή μας. Όλα αυτά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι γίνονται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε. Η, η κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη εμφανίζονται στο τιμίο που αναφέρονται οι τομείς Αρμοδιότητα ε, πολιτικής συνοχής. Εκεί φαίνονται όλες οι αρμοδιότητες που εμπίπτουν ε, στον τομέα των ε, κρατών μελών. Έντις. Το Έντις είναι ένας νέος φορέας που πρωτοεισήχθη με τον προϋπολογισμό του 2019 Ανταποκρινόμενοι και σε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ακόμα βρίσκεται στο στάδιο της ε, προετοιμασίας. Η η υπηρεσία μα, οι μας ε, ακόμη εκπαιδεύονται, ξέρετε. Οπότε ε, ο αριθμός αυτός των ε, ε, των ε, περιπτώσεων 6 που αναφέρατε θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Γιατί χρειαζόμαστε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον όλο αυτόν έχουμε εδώ και δεκαετίες. Όλαφ διερευνά περιπτώσεις απάτης και παρατυπίες. Η απάτη, λοιπόν, όμως ρυθμίζεται νομοθετικά σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για περιπτώσεις κατάχρησης χρημάτων κάποιου άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου ε, εμπροκειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μπορεί να υπάρξουν διάφορες μορφές, λάθος αριθμητικά στοιχεία ή και μη σκόπιμες ε, παρατυπίες, οι οποίες όμως παρόλα αυτά εξακολουθούν να είναι μη αποδεκτές. Στο Διεθνέ ποινικό δίκαιο υπάρχει συμφωνία για το πώς μπορεί κανείς να ορίσει τα ζητήματα της απάτης, της διαφθοράς και της παρατυπίας. Παρ' όλα αυτά το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται νομοθετικά σε εθνικό επίπεδο και έτσι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το ποινικό δίκαιο είναι εθνική αρμοδιότητα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είχαμε λοιπόν μέχρι σήμερα μια ποινική υπόθεση, μια απάτη, ένα φυσικό πρόσωπο ε, ε, βρίσκεται υπό διερεύνηση και καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ότι, υπάρξει, ότι έχει υπάρξει απάτη αυτού του μεγέθους, αυτής της έκτασης. Σε, εκεί τελειώνει και το, το, έργο μας. Μπορούμε να ανακτήσουμε τα χρήματα ώστε να εισπραχθούν υπέρ του ευρωπαϊκού ε, προπολογισμού, αλλά από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι εθνικέ αρχέ. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν πολύ μεγάλε διαφορέ όσον αφορά την προθυμία να προχωρήσουν αυτέ οι υποθέσει. Γι' αυτό και επιδιώξαμε να υπάρξει ένα εναρμονισμένο τρόπο Αντιμετώπιση αυτών των υποθέσεων και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο Όλαφ θα μπορεί να παραδίδει αυτές τι υποθέσεις στην ε, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορεί να προσφεύγει στα εθνικά δικαστήρια με πρότυπα και κανόνε που θα είναι ενιαίοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα συνεκτικότερο επίπεδο δικαιοσύνη αν θέλετε, σε σχέση με το παρελθόν. Μπορούμε να πούμε ότι όλα είναι η αστυνομία και η ΕΠΟ είναι η εισαγγελία. Η αστυνομία είναι εκείνη που πηγαίνει σε μια διάρρηξη, παίρνει δακτυλικά αποτελέσματα, συλλέγει τα στοιχεία, τα πηγαίνει μετά στην εισαγγελία, η οποία στη συνέχεια ε, εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου. Δεν έχουμε ακόμη ποινικό δικαστήριο ευρωπαϊκό. Ίσως θα μπορούσε να είναι ένα επόμενο βήμα. Όμως, στον τομέα του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού και των ε, περιπτώσεων απάτης εις βάρος του, ο Όλαφ συγκεντρώνει τα στοιχεία, από εκεί και πέρα ε, παραδίδει αυτά τα στοιχεία αυτά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα μπορούσε ε, κάποια στιγμή να προβλεφθεί να συσταθεί και ένα Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο. Το αν θα επιλεγεί μια τέτοια προοπτική δεν σε μένα να το πω, όμως είναι, σας περιγράφω τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαμορφώσει την καταπολέμηση της απάτης. Προστασία ε, δεδομένων και διαφάνεια. Εμείς στηρούμε απαρέγκλητα τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και θα ήθελα να πω ότι και ε, ε, σε ερωτήσεις, λόγω των ερωτήσεων των Ευρωβουλευτών, εμείς είμαστε πάντοτε υποχρεωμένοι να τηρούμε τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πολλές φορές δηλαδή εσείς οι ίδιοι μας καλείτε ε, να προστατεύουμε τα, προσωπικά δεδομένα. Όμως, ωστόσο, όταν μια υπόθεση ερευνάται δικαστικά, τότε τα πράγματα είναι δημόσια. Εκεί βεβαίω τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κανονικά κάναμε λάθο. Πρώτα ακούμε του ε, εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια τον ε, εισηγητή. Κάναμε, έκανα αυτό το λάθο, αλλά εν πάση περιπτώσει α δώσουμε τώρα τον ε, λόγο στου συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Σα ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Επίτροπε, σα ευχαριστούμε πολύ και την Επιτροπή γενικά για την έκθεση αυτή. Και εδώ βλέπουμε μια σύνοψη τη δραστηριότητα τη τελευταία πενταετία, όχι τρία κονταετία, και βλέπουμε την εισαγγελία, την ε, πύφη για τα οικονομικά συμφέροντα, το Όλαφ, τη στρατηγική, όλα αυτά πολύ σημαντικά για την τελευταία πενταετία. Από την άλλη πλευρά όμως δυστυχώς η ίδια Επιτροπή έκανε την έκθεση την ε, διετή ε, και είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο Μπαρόσο και το λόμπι που έκανε και το ότι πήρε τη θεσούλα στο Goldman Sachs και τι έγινε επίσης και με το Γενικό Γραμματεία της Κομισιόν αυτά δυσαρ... όντως έχω τις εξής παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα, η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΠΙΦ ήταν Ιούλιος του 19. Θα πρέπει να κάνει την αξιολόγηση η Κομισιόν μέχρι το 2021 για την ε, ε, θέσπιση τέλο πάντων εφαρμογή τη οδηγία. Τι γίνεται, πόσα κρατημέλη το κάνανε, πόσα δεν το κάνανε, πόσα έβαλαν στην ένωμη του στην ε, οδηγία, ε, εμπρόθεσμα. Επίσης λέτε να τροποποιηθεί ο 883 ο κανονισμό για την Όλαφ και έτσι να προσαρμοστεί η λειτουργία της Όλαφ. Όμως δεν άρχισαν να όφυλαν οι διαπραγματεύσει. Άρα θα αργήσει η θέψη του κανονισμού ω όφιλε. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να γίνει αρχή της χρονιάς. Τι γίνεται. Η ΕΠΟ είναι ε, ήδη επιχειρησιακή, ήδη λειτουργεί τέλο πάντων, αλλά δεν υπάρχει ο κανονισμός που πρέπει τελευταίο. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπόσχεται να καταπολεμήσει τις απάτες, αλλά δεν έχουν γίνει οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει να μπείτε στο συνθήκη Γκρέκο. Σα παρακαλώ. Παρακαλώ όλους του συναδέλφου. Σας παρακαλώ, αν θέλουμε να μα παίρνουν σοβαρά στην κόλ. Καλό είναι να ακούμε γενικά απόψεις, αλλά λοιπόν σας παρακαλώ να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε ορισμένα άτομα για απάτες. Και για τον κύριο Μπαρόζο και για τον κύριο Ζελμάιερ. Μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε προσωπική γνώμη για το τι έκαναν, αλλά να λέτε ότι συνδέεται ο διορισμός τους, ο οποίος ελέγχθηκε νομικά πριν εγκριθεί με περιπτώσεις απάτης. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο κύριος Δένας που είναι σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λίγο απογοητεύτηκα. Είμαι σχετικά καινούριο εδώ και για λίγο θεώρησα ότι όλοι θα μιλάμε τον ίδιο χρόνο. Όπως και ο Επίτροπος. Αυτό θα ήταν πολύ γενναιόδωρο. Οπότε ετοίμασε ομιλία 15 λεπτό και τώρα πάει. Μου λέτε για 1,5 λεπτό. Καλά θα προσπαθήσω. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο και την Όλαφ για την έκθεση του περασμένου μήνα. Είναι εξαιρετική η έκθεση, ιδίω όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση. Το θέμα είναι ένα από τα θέματα και θα πρέπει να τα πούμε ότι δεν σημαίνει και πολλά εν προκειμένου η ανάλυση. Τα λέει η ίδια η Επιτροπή ότι τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν πόσες περιπτώσεις ε, εν δυνάμει απάτης αναφέρονται από τα κράτη-μέλη, όμως στην πραγματικότητα, στην πράξη, πόσες απάτες είχαμε. Κάνουμε κάθε χρόνο τέτοιες ε, εκθέσεις και θα πρέπει να πούμε κάτι λογικό. Αυξάνεται, μειώνεται, τα πάμε καλύτερα στην αντιμετώπιση. Ξέρω ότι τον Απρίλιο βγήκε, αλλά αυτή η στρατηγική κατά τις απάτες της Κομισιόν βοηθάει όσον αφορά αυτή την ε, πλευρά σε σχέση με την ανάλυση. Και κάτι άλλο. Αναφέρεται στην έκθεση την πρόταση της Κομισιόν για προστασία του προϋπολογισμού, του κράτους δικαίου Μόνο 11 κράτη-μέλη έχουν στρατηγικές κατά τις απάτες μέχρι τώρα. Ελπίζουμε ότι και άλλες θα κάνουν το ίδιο, αλλά εσείς η εθνική τέτοια στρατηγική θα βοηθήσει στο να πληρούνται αυτή η προϋπόθεση του κράτους δικαίου για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις πολύ συγκεκριμένες και πραγματικά επικοδομικές ερωτήσεις. Παρακαλώ η Κατρίνα Κινίτση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο για όσα μας παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή. Μας τόνισε ότι εδώ και 30 χρόνια καταβούμε την απάτη και έχουμε ένα σωρό βελτιώσει αυτή την 30 ετία. Πάντως, πάντοτε αναδύονται καινούργιε προκλήσει, όπω την περσμένη εβδομάδα στην Επιτροπή που μιλήσαμε για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι σημαντική η καινοτομία για τον κόσμο, αλλά, αλλά μας ε, δείχνει ε, ακόμα μια πλευρά απάτες ιδίω όσον αφορά τα τελωνιακά. Οπότε γίνεται τώρα η προσπάθεια τα υπόλοιπα οι 22 κράτη της ενσυμμένης εργασίας να μπορέσουν να προσχωρήσουν ε, στα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συμφωνώ ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά τον κανονισμό της ε, Όλαφ για να μπορέσει και η Όλαφ και η Εισαγγελία να χρησιμοποιηθούν ως σημαντικό μέσο κατά τις ε, απάτες και όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Μια γενική ειδική ερώτηση. Θα πρέπει πιο συγκεκριμένα να δούμε αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε. Γιατί, για να είναι αποτελεσματική προστασία των νομικών συμφερόντων, θα πρέπει να υπάρχει ε, ομοιογένεια όσον αφορά την νομοθεσία και τις ε, επεμβάσεις μας. Και οι εθνικές ε, αρχές θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με αυτές τις δόλειες και μη ε, ε, λήψει και παρατυπίες, οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πρακτική σήμερα σχετικά με αυτόν τον κρατών μέλλον. Ορισμός της απάτης και παρατυπίες και συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά μας απασχολούν εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι κάτι το νέο, όλα αυτά είναι παγιωμένα. Οπότε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα υπάρχει περισσότερη ομοιογένεια από πρακτικής πλευράς, από επιχειρηματική πλευράς όσον αφορά την επισήμανση των παρατυπιών από και για τις εθνικές αρχές. Πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε αποτελεσματικά να, αποτελε... να... καταπολεμήσουμε το έγκλημα και τις παρατυπίες ει βάρο των οικονομικών συμφερόντων της ενωση πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στρουγκάριο. Thank you so much. Um... Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, για το Renew είμαστε οι σκιώδεις εισηγητές, οπότε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Τροπή για όσα έκανε σε αυτή την έκθεση και γενικότερα για το έργο της σε αυτό το μέτωπο. Το 2019 έχουμε κλείσει 30 χρόνια όσον αφορά τις προσπάθειες για προστασία των οικονομικών συμφερόντων και σε αυτά τα 30 χρόνια Έχουμε κάνει πολλά, πολλές ε, προκλήσεις, άλλαξαν μορφή. Θα πρέπει να υπάρξει εξασφάλιση της, ε, των οικονομικών συμφέροντων περισσότερο. Οπότε τώρα για να δούμε κάποια από αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος ε, εισηγητής. Να δούμε μερικά στοιχεία. Πολύ ανησυχητικό ότι σε σχέση με το 17 παρά το ότι οι δόλειες παρατυπίες ελαφρώς μειώθηκαν ή μείναν ίδιες αυξήθηκε κατά 183% το σχετικό αριθμητικό ποσό. Αυτό σημαίνει με ένα μεγάλο χτύπημα στον προπολογισμό. Επίσης, είχαμε μεγάλη χρηματοδότηση σε τομεί όπως τη Γεωργία, αλλά οι παρατυπίες από δύο κρατημέλη, Ρουμανία και Ιταλία, είναι άνω του 60% όλων των παρατυπιών της Ένωσης, το 19%. Η Ρουμανία είναι πρωταθλήτρια εδώ η χώρα μου. Καλά, να μην είμαι τώρα εθνικήστρια ούτε λαϊκήστρια. Ε, γιατί έτσι θα είμαι πατριώτης, άμα σας πω την αλήθεια. Ουγγαρία και Πολωνία επίσης είναι δύο από τα έξι κρατημέλη που δεν έχουν μπει στην εισαγγελία και εκεί ε, υπάρχει επίκληση του άρθρου 7 εις βάρος τους, όσον αφορά το κράτος δικαίου τώρα. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε γιατί αλλιώ αλλιώς υπάρχει απειλή για τον προϋπολογισμό η εισαγγελία είναι μεγάλο βήμα για προστασία των συμφερόντων της Ένωσης. Όμως, α, ακόμα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που μας περιμένουν και πρώτα-πρώτα το πώς όλα τα κρατημέλη θα προσχωρήσουν. Δεύτερον, θα πρέπει εδώ να δουλέψουμε σωστά, καλύτερη παρακολούθηση και αποτελεσματικές κυρώσεις. Έτσι θα πετύχουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων. Τρίτο και σημαντικό, και τα κρατη θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο. Θα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα κατά τις απάτες και εθνικές στρατηγικές, γιατί προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σημαίνει προστασία των οικονομικών του κάθε πολίτη χωριστά, του κάθε Ευρωπαίου. Και για αυτό και χρειαζόμαστε τέτοια μέσα πολιτική σε επίπεδο Ένωσης. Διακόπτη η Πρόεδρος. Τρία λεπτά, τρία λεπτά μιλήσατε ήδη, τη λέει. Ευχαριστώ. Σαρβαμά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την έκθεση, την ανάλυση, τις συστάσεις σας και η εμπειρογνωμοσύνη της Όλαφ για την απάτη είναι κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει πολύ. Πέραν αυτού τώρα συμφωνώ με, την σκιώδη, με τον σκιώδη, σκιώδη τον κύριο Λέναρς. Δυστυχώς. Εδώ κάνουμε κάτι σαν λογιστική. Δεν κατανοούμε τι πραγματικά συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Πάντως, εντάξει, δεν λέω ότι φταίει για αυτό ούτε η Επιτροπή, ούτε ο Επίτροπος. Αλλά τελικά, αν δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε όλο το τοπίο και τις μεταβολές του, δεν φτάνουν τα αριθμητικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Τέλος. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Έτιγκερ, από καρδιάς για τα όσα κάνατε αυτή την ε, πενταετία που ήταν πολύ αξιόλογα. Ευχαριστούμε για την άγαστη συνεργασία επίσης. Vielen Dank, γερμανικά. Λοιπόν, θα είχα και εγώ μία ερώτηση προς τον Επίτροπο. Διότι υπάρχουν όλο και πιο περίεργες διαδικασίες, πιο πονηρές διαδικασίες. Έχετε νέους τρόπους αντιμετώπισης. Κοιτάξτε. Μπορεί να αξίζει το κόπο να κάνεις απάτη. Γιατί έχει κάνει τον υπολογισμό του. Δηλαδή, τι πιθανότητα υπάρχει να βγάλω κάποια λεφτά και τι θα μου κοστίσει Άρα τελικά μπορεί να με συμφέρει ακόμη και αν με πιάσουν. Και αυτό δημιουργεί βέβαια στρεβλό στην αγορά. Έχετε αποκαλύψει, έχετε ανακαλύψει όλο και περισσότερο νέα τέτοια συστήματα. Υπάρχει μια περίπτωση που μπορείτε να μας ε, περιγράψετε. Και οι ποινές είναι τόσο υψηλές, όντως, ούτως ώστε ε, να μην έχει κέρδος όποιος το επιχειρεί. Λοιπόν, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Για την τελευταία ερώτηση. Αν ε, οι επιπτώσεις μιας απάτης και αν ε, ο απατεώνας μπορεί να κάνει μια αποτίμηση κόστους, ωφέλους. Εάν αποκαλύψουμε μια απάτη. Δεν μένει τίποτα στον ε, διαπράξαντα στο τέλος και επιπλέον βέβαια ε, μετά υπάρχει και ποινή η οποία βέβαια εξαρτάται από το εθνικό δίκαιο. Οι απάτη και οι σοβαρές απάτες μπορεί να έχουν σε επίπτωση πρόστιμα αλλά και ποινές φυλάκισης. Αυτό είναι και συνεχίζει να είναι πλήρης ευθύνη του εθνικού νομοθέτη. Στην έκθεσή μας έχουμε διαπιστώσει όλο και πιο πονηρές και περίπλοκες ε, περιπτώσεις απάτης. Και εκεί δείχνουμε προς τα που πάνε οι εξελίξεις. Για παράδειγμα, ηλεκτρονικό εμπόριο. Και γενικά στο ψηφιακό κλάδο αλλάζουν οι μέθοδοι. Οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν βέβαια πολλά θετικά, αλλά ε, περιέχουν και κινδύνους. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν υπάρξει διάφορες ανισχυτικές εξελίξεις αλλά προσπαθούμε να, τις, ε, να προσαρμόσουμε την εργασία μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κόλπα που είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Εάν αυξάνεται το ποσό των απατών, συνήθως αυτό έχει με μία-δύο περιπτώσεις ε, απατών υψηλού επίπεδου. Γιατί ξέρετε, ξέρετε, οι περιπτώσει είναι περίπου οι ίδιε, αλλά μετά έρχεται μια χοντρή περίπτωση και αυξάνει κατά πολύ το ποσό που εμπλέκεται στι απάτε. Και μετά την επόμενη χρονιά πέφτει πάλι. Η σύσταση για να υπάρξει εθνική στρατηγική καταπολέμηση των απατών είναι ακριβώ αυτό μια σύσταση. Δεν έχω κανένα περίστροφο για να το θέσω στο κρόταφο των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων. Αλλά ορισμένοι που μιλήσανε είναι ακριβώς από τα κράτη-μέλη που ε, ακριβώς σημειώνονται οι απάτες. Ε, οπότε εσείς έχετε πολύ περισσότερες. Κοιτάξτε, είναι σαν να είστε εσείς στο Κολοσσέο στο θεωρείο του αυτοκράτορα και εγώ είμαι κάτω στην αρένα και μου επιτίθενται τα λιοντάρια που τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Στην Πράγα, στο Βουδαπέ, στο Βερολίνο, τη Ρώμη, το Βουκουρέστι, τη Σόφια. Δεν μπορούμε να πετάξουμε και με το πολυβόλο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συγκεντρωτικό κράτος. Και το Κοινοβούλιο και εμείς έχουμε περιορισμένες δυνατότητες δράσης. Αλλά αν δείτε τι γινόταν στο παρελθόν, έχουμε επιτύχει πολλά. Πριν από 20 χρόνια, ο οργανισμός Όλαφ ε, δεν είχε τις δυνατότητες που έχει σήμερα. Πριν από 20 χρόνια τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θεωρούσαν μια γραμματεία για να διεκπαιρώνουν τις υποθέσεις τους. Όσο προχωράμε μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλο και περισσότερο τις προσδοκίες σας. Για την εφαρμογή της οδηγίας PIF. 12 κράτη-μέλη την έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο. 8 την έχουν μεταφέρει εν μέρη και τα υπόλοιπα καθόλου. Τι μας μένει. Μας μένει να κάνουμε προσφυγή επί παραβάση. Και θα το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα βέβαια κάνουμε συζήτηση, μετά κάνουμε εκκλήσεις, αλλά και στο τέλος μπορεί να υπάρξει και νομική διαδικασία. Να απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και, κοιτάξτε, ε, πολύ φιλικά, οι περιπτώσεις Μπαρόζο και Ζελ δεν έχει ε, καμία σχέση με απάτε. Έχουν γραφτεί διάφορες βλακίε στον τύπο. Κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα διοικητικού δικαίου, αλλά απάτη, καμία σχέση. Μπορούμε να, να θέσουμε θέματα δεοντολογίας, αλλά όχι, όχι. Δεν είναι η σωστή στιγμή και ο σωστό χώρο και το σωστό όργανο για να λέτε τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να δυσφημούνται συνάδελφοι που μπορεί να είναι ε, συζητήσιμη συμπεριφορά τους αλλά δεν έχουν καμία σχέση με απάτες. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Θέλω στο τέλος να ευχαριστήσω προσωπικά ως πρόεδρος την, τον Επίτροπο γιατί τα τελευταία χρόνια η συνεργασία μεταξύ του Επιτρόπου και της Επιτροπής Ελέγχου του Ευρωπαϊκού ήταν ε, εξαιρετική και εκφράζω την άποψη αυτή και εξ ονόματος εκείνων που κατήχαν τη δική μου θέση καθόλου τη, διάρκεια αυτής της τριετίας. Σας ε, ευχόμαστε, ευχόμαστε μάλλον, αυτά που ξεκινήσατε εσείς ε, να τα συνεχίσουμε εμείς εδώ από το μετερίζι της Κοντ και να βασιστούμε σε αυτά και στο μελλοντικό μας ε, έργο. Να δώσω λόγο το λόγο ξανά στον κύριο Κούς ως εισηγητή. Θέλω πάντως ε, να ευχαριστήσω τον κύριο Έτιγκερ ε, για την ε, εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ο Ιωάννης Χάν βεβαίως μια χαρά θα είναι και εκείνος, αλλά σχεδόν συγκινούμε, κύριε Έτιγκερ, που σας αποχαιρετώ. Κύριε Κούς, παρακαλώ. Genau. Ich möchte mich den ε, να συμφωνήσω και εγώ και να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Έτιγκερ. Ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισα. Ε, που σχημάτισα από εσάς έχω πιστεί ότι πραγματικά είστε πάντοτε πολύ ενδελεχείς στις απαντήσεις σας, πολύ προσεκτικός. Ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε και με τον επόμενο επίτροπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι. Kommen nun zu Tagesordnungspunkt. Περνάμε στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Να σας παρακαλέσω να καθίσετε σας παρακαλώ και να σταματήσουν οι ομιλίες αν γίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα Καταρχάς, να καλωσορίσω τον κύριο Νικόλα, Νικόλα που είναι τα, και τα υπόλοιπα αρμόδια μέλη του ε, Ευρω... Ε, Ελεγκτικού Συνεδρίου και θέλω να ευχαριστήσω παρά τη γρήπη ότι ήρθε εδώ και είναι μαζί μας ο Επίτροπος. Ξέρω ότι βρίσκεται σε έξαρση. Θέλω να δώσω λοιπόν ε, τον λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο και στη συνέχεια θα δώσουμε βέβαια το λόγο και στον Επίτροπο για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να σας ε, παρουσιάσω τη δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με, την, ε, με τον τομέα 2, φυσική πόρη. Για το 2018 το ποσοστό σφάλματος εκτιμάται στο 2,4% για τον τομέα φυσική πόρη συνολικά είναι παρόμοιο ε, το ποσοστό αυτό με τα όσα είχαμε εντοπίσει τα δύο, προγραμμα... Ε, τα προηγούμενα χρόνια και πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2%. Οι σύνθετοι όροι επιλεξιμότητας ε, είναι αυτοί που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ασφάλματος. Στις δαπάνες που ελέγξαμε εμείς περιλαμβάνεται η αγροτική ανάπτυξη, ε, τα μέτρα στήριξης αγοράς, ε, αλληλεία, περιβάλλον. Από τις 156 πληρωμέ που ελέγξαμε σε αυτού του τομείς ψηλού κινδύνου, ένα τέταρτο περίπου ε, εμφάνιζαν σφάλματα. Οι βασικοί λόγοι σφάλματος σχετίζονταν με τους όρους επιλεξιμότητας, τους κανόνες δημοσίων συμβάσεων και επιχορηγήσεων και ανακριβείς ε, πληροφορίες όσον αφορά τι εκτάσει. Για παράδειγμα, βρήκαμε ένα δικαιούχο που, δικαιούχο που η εκμετάλλευσή του η, εκμετάλλευσή του ήταν πολύ μεγάλη για να λάβει την στήριξη που λάμβανε. Ή άλλος ε, εμφανιζόταν ως νέος γεωργός, ενώ ε, ήταν την πρώτη χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα σταμάτησε να πληρεί τον, τον όρο για τους νέους γεωργούς. Πέρσι συστήσαμε στην Κομισιόν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δράσεων των κρατών μελών για να αντιμετωπιστούν οι αιτίε των σφαλμάτων και να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές όπου χρειαζόταν. Αυτή η ανοιχτή σύσταση ισχύει και για τα όσα βρήκαμε το 2018. Θα αξιολογήσουμε την ε, εφαρμογή αυτή στο πλαίσιο των από εδώ και πέρα εργασιών μας. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα του προπολογισμού αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις του Ταμείου Εγγυήσεων. Ε, εδώ εκτιμήσαμε το ποσοστό σφάλματος να είναι κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2%. Αυτό επιβεβαιώνει τα, τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε βρει και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Από τις 95 ε, άμεσες ενισχύσεις που ελέγξαμε, 81% δεν εμφάνιζαν σφάλμα και τα περισσότερα σφάλματα που βρήκαμε ήταν μικρέ ε, υπερ, ε, ε, υπερπληρωμές κάτω από 5% λόγω κυρίως γεωργών που μας έδιναν ανακριβείς πληροφορίες για τις εκτάσεις τους. Τα θετικά επιτεύγματα όσον αφορά τι άμεσε ενισχύσει του Ταμείου Εγγυήσεων οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση και ελέγχου, το Ajax, το σύστημα εντοπισμού ε, αγροτεμαχίων και την εφαρμογή γεωχωρικής βοήθειας καθώς και τους ε, διασταυρούμενους ελέγχους που διενεργούνται στις αιτήσει των γεωργών. Στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και ε, επιδόσεων 2018 η Κομισιόν παρουσιάζει επίπεδα σφάλματος 2,1% για τις δαπάνες της κοινή γεωργικής πολιτικής στο σύνολο και 1,8% για τις άμεσες ενισχύσεις των μειογγύσεων. Αυτά τα στοιχεία ε, συμφωνούν και με τα δικά μας συμπεράσματα των ελέγχων ότι το επίπεδο του σφάλματος στους φυσικούς πόρους ήταν σημαντικό ενώ στις άμεσες ενισχύσεις ε, δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το ποσοστό σφάλματος. Από το 2015, οι φορείς πιστοποίηση είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με την νομιμότητα και την ε, τυπικότητα των δαπανών για, τα, για τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει επιστροφές. Το 2018, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, πραγματοποίησε... Ε, επισκέψεις σε 17 φορείς πιστοποίησης και μόνο από 5 από αυτούς φάνηκε ότι είναι αξιόπιστοι. Προσδιορίσε η DG Agri διάφορα ζητήματα όσον αφορά την ε, μεθοδολογία δειγματοληψίας και τους ελέγχους επιλεξιμότητας. Και η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, στην έκδοση των δικών της επιπέδων σφαλμάτων για, την, για τις δαπάνες ΚΑΠ έκανε κάποιες προσαρμογές. Λαμβάνοντα υπόψη τους, ε, τα στατιστικά στοιχεία ελέγχου των ε, οργανισμών πληρωμών. Όπω και τα προηγούμενα χρόνια, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας βάσισε τι περισσότερε προσαρμογέ της στους δικούς της ε, ελέγχους συμμόρφωση των δαπανών των οργανισμών πληρωμών. Όμως για να υπάρξει συνεχής και ε, συνεκτική βελτίωση χρειάζεται η Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι και τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί είναι πραγματικά αξιόπιστα. Το 2018 επίσης εκδώσαμε ένα ενημερωτικό έγγραφο για, την, για το μέλλον της ΚΑΠ και μια γνωμοδότηση για τις νομοθετικές προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2020. Όσον αφορά τις επιδόσεις, Έχουμε εκδώσει ε, πρόσφατα και κάποιες ειδικέ εκθέσεις για ζητήματα που σχετίζονται με την κοινή γεωργική πολιτική, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το βασικό καθεστώς ενισχύσεων, τις επιλογές απλοποιημένου κόστος για την χρηματοδότηση έργων αγροτικής ανάπτυξης και ευζοίας των ζώων. Επίσης, καλύψαμε περιβαλλοντικά θέματα, ιδίως τη ρήπανση του αέρα, την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, την αντιπλημμυρική προστασία και την ερημοποίηση. Οι επισκέψεις μας σε δικαιούχου για τη δήλωση αξιοπιστίας ήταν επίσης και μια ευκαιρία για να ε, αξιολογήσουμε και τα στοιχεία των επιδόσεων. Βρήκαμε ότι οι δράσεις αγροτικής ανάπτυξης γενικά είχαν διεξαχθεί όπως είχαν σχεδιαστεί και ότι ε, ήταν εύλογο το κόστος τους. Είχαμε στο παρελθόν επισημάνει ότι για κάποια έργα οι επιλογές απλοποιημένου κόστο όπω. η καταποκοπή ποσά ή τα καταποκοπή ποσοστά έχουν τη δυνατότητα να απλοποιήσουν την, ε, τον διοικητικό φόρτο και να τηρούν σε ελέγξιμα επίπεδα το κόστος. Και αυτό ε, ισχύει ιδίως για μέτρα που περιλαμβάνουν δράσεις με παρόμοιους το, τύπους δραστηριοτήτων και δαπανών. Και βρήκαμε ότι οι εθνικές αρχές σε πολύ μικρό βαθμό χρησιμοποίησαν αυτές τις ε, επιλογές ε, απλοποιημένου κόστους, αν και θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Εξετάσαμε και την, ε, το πλαίσιο που χρησιμοποιεί η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για τη μέτρηση των ε, επιδόσεων και την υποβολή εκθέσεων υπό την ΚΑΠ. Και διαπιστώσαμε ότι περίπου το 1 τρίτο από τις δράσεις των αγροτικών, ε, ε, αγροτικής ανάπτυξης δεν είχαν κάποιον δίκτυ αποτέλεσμα, αποτελέσματος. και στις μισές από αυτές τι περιπτώσεις αυτοί οι δείκτες ορίζονταν βεβαίως σε εθνικό επίπεδο. Όπου ε, ορίζονταν, πολλέ πολλές φορές αυτοί οι δείκτες όμως δεν σχετίζονταν με τους στόχους των ε, τομέων επικέντρωσης προσοχής. Γι' αυτό και εμείς ε, συστήσαμε η Κομισιόν να άρει αυτές τις αδυναμίες στο πλαίσιο τη πρόταση που θα υποβάλει για την νέα κοινή γεωργική πολιτική. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιλιώνη. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χόγκαν τώρα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ε, ως Προέδρο αυτής της σημαντικής επιτροπής. Και είναι η έκτη φορά που έρχομαι για να συζητήσουμε τη διαχείριση και την απόδοση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι η τελευταία φορά όμως που θα εμφανιστώ ενώπιόν σας ε, υπ' αυτήν την ιδιότητα και ξέρω πόσο σημαντική είναι αυτή η αιτήσια ανταλλαγή απόψεων και τι δυνατότητες μας δίνει. Φυσικά είναι πολύ σημαντική η επίβλεψή σας για να υπάρχει δημόσια εμπιστοσύνη και ένα ρωμαλαίο σύστημα για να προστατεύσουμε τη δαπάνηση των δημοσίων πόρων και για να μπορούν όλοι οι επίτροποι να λογοδοτούν. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την απαλλαγή του 2018 και θα ασχοληθούμε με αυτήν και τα τελευταία πέντε χρόνια. Η κοινή γεωργική πολιτική και φέτο έδωσε προστιθέμενη αξία για του Ευρωπαίου πολίτε. Οι δαπάνε τη ε, είναι σωστέ και βασίζονται, πληρούν μάλλον, τα κριτήρια. Έχουμε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ε, ε, ε Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Η αξιοπιστία μα είναι στο 98,5% και το συνέδριο καταλήγει σε παρόμοια ε, πορίσματα. Για τους φυσικούς πόρους το συνέδριο λέει ότι τα σφάλματα είναι 2,4% το οποίο είναι παρόμοιο και με άλλους τομείς. Ενώ η Κομισιόν λέει ότι είναι στο 2,15. Επιπλέον υπάρχουν πολλά μερικά θετικά μηνύματα από το συνέδριο και από την ετήσια αυτή έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Οι άμεσες πληρωμές και φέτος δεν έχουν ουσιώδη λάθη το συνολικό ποσοστό είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σφαλμάτων δηλαδή. Και έχει βελτιωθεί η εργασία των οργανισμών πιστοποίησης. Αυτή η θετική άποψη του συνεδρίου αντανακλάται και στο γεγονό ότι φέτος δεν μας κάνουν ε, συστάσεις για βελτίωση της αξιοπιστίας σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική. Και αυτό οπωσδήποτε δείχνει ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν κάνει σκληρή δουλειά. Τα κράτη-μέλη κάνουν σκληρή δουλειά για να γίνεται σωστά η εκταμείευση των πόρων. Και επίση και η Κομισιόν για να εντοπίσει τα λάθη και να προτείνει συστημικέ λύσει. Με βάση με τι συμβουλέ που έχει δώσει η Επιτροπή σα και βεβαίω ε, ε, τι συμβουλέ των κρατών μελών. Και τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να βελτιώσουν τα συστήματά του και αυτά έχουν θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, καλωσορίζω το γεγονό ότι το συνέδριο στην έκθεσή του επιβεβαιώνει ότι το σύστημα εντοπισμού των αγροτοτεμαχίων συμβάλλει ιδιαίτερα στη μείωση του επίπεδου λαθών. Φυσικά, το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την κατάσταση των ε, πληρωμών που βασίζονται ε, στις ε, επιφάνειες. Όμως το σύστημα των άλλων επιδοτήσεων για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι πιο περίπλοκο. Παρά την περιπλοκότητα όμως έχουμε επιτύχει πολλά. Έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές από τις αδυναμίες. Οι πρωτοβουλίε που έχουμε αναλάβει αρχίζουν να αποδίδουν. Απλουστεύσαμε και βελτιώσαμε την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Τα κράτη-μέλη έχουν προγράμματα δράσης που τα εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα αρχίζουν και φαίνονται. Αυτό ε, αντανακλάται και στο ποσοστό σφαλμάτων. Κυρία Πρόεδρε, κάποιες ανησυχίες που έχουν να κάνουν με κάποιες περιπτώσεις απατών και σύγκρουση συμφερόντων που έχουν περάσει και στον τύπο. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή και η Ανεξάρτητη Όλαφ ασχολείται πολύ σοβαρά με τα θέματα αυτά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προστατεύσουμε τον προπολογισμό τη Ένωση και θα αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε, του κανονισμού. Κάθε υποψία απατών και σύγκρουση συμφερόντων που θα ε, υποπέσει στην αντίληψή μα θα αντιμετωπιστεί κατάλληλα, θα ληφθούν τα μέτρα για να ε, προστατευτεί ο προπολογισμό τη Ένωση. Αυτέ οι λίγε περιπτώσει δεν θα πρέπει να μα επιτρέψουν να αμαυρωθεί η εικόνα των δαπανών που, για την κοινή γεωρική πολιτική που είναι σωστή. Υπάρχει λοιπόν υψηλή αξιοπιστία για τι δαπάνε τη ε, κοινή γεωργικής πολιτική. Τα σφάλματα είναι κάτω από το επίπεδο σημαντικότητα. Και έχουμε και ένα ρωμαλαίο σύστημα διορθωτικών ενεργειών που εφαρμόζονται όταν είναι αναγκαίο. Και αν αφαιρέσουμε τι ε, διορθώσεις και αυτά που παίρνουμε πίσω από του δικαιούχου, το ποσοστό που παγωμένει είναι 0,25. Αυτό σημαίνει ότι δαπανούμε σωστά τα χρήματα. Η εφαρμογή τη ε, κοινή γεωργική πολιτική και του προπολογισμού τη και οι άμεσες πληρωμές έχουν θαυμάσιο ποσοστό απορρόφηση. Περίπου 99% των πόρων απορροφήθηκαν το 2018. Και για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου έχουμε νέα προγράμματα. Το 38% έχει διπληρωθεί. Είναι 47,7 ε, δις. Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε μια καλή δομή διακυβέρνηση για την ε, κοινή γεωρική πολιτική και τώρα θα μιλήσουμε για την απόδοση. Τι γίνεται λοιπόν τώρα από πλευράς της απόδοσης. Και το βασικό είναι να υπάρχουν θέσει απασχόληση στη Γεωργία. Η Γεωργία είναι η κύρια δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Πάνω από 44 εκατομμύρια εργαζόμενοι εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα στον άγρι διατροφικό τομέα. Είναι όμως ευάλωτος αυτός ο τομέας. Χρειάζεται προστασία από τις πιέσεις ε, των αγορών. Άρα στηρίζω τι άμεσε πληρωμέ, τη συνέχιση τους. Ε, ξέρω ότι αυτό προκαλεί κάποιε συζητήσει, αλλά είναι μια βάση εισοδήματο. Είναι ένα βασικό εισόδημα για του γεωργού μα και μια πηγή σταθερότητα για την εργασία του. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε και το περιβάλλον. Οι πληρωμές πρέπει να έχουν να κάνουν και με την προστασία του περιβάλλοντο. Γίνονται κάποιε κριτικέ κάποιε επικρίσεις για τη διανομή των άμεσων πληρωμών. Δεν δικαιολογείται. Αυτό το αποδεικνύουν οι πρόσφατε μελέτε. 72% των βοηθειών αυτών πληρώνεται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις μεταξύ 5 και 250 εκταρίων. Οι μισοί δικαιούχοι έχουν λιγότερο από 5 εκτάρια. Αυτό αποδεικνύει ότι το σύστημα πραγματικά δεν αφήνει κανένα στο περιθώριο. Και περιέχει και την υποχρεωτική ε, πτωτική τάση των πληρωμών όσο αυξάνεται η επιφάνεια και ένα σύστημα αναδιανομής. Φυσικά μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις, αλλά αυτό το προτείνω. Κάνω προτάσεις για μετά το 2020 για και ανώτατα όρια και ένα σύστημα που θα μειώνει τις αμοιβέ όσο αυξάνεται η επιφάνεια. Αυτό ισχύει στη Γερμανία ήδη. Έχουμε δώσει πολλές πληρωμές για την αναδιάρθρωση και έχουμε στηρίξει 106.000 νέων γεωργών για να δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους. Έχουμε αυξήσει το ποσοστό αυτό ε, λοιπόν πολύ και έχουμε αυξήσει και το ποσοστό από 11 σε 53% μεταξύ 2011 και 2018 για να υπάρξει ευρυζωνική σύνδεση παντού στην Ήπεθρο. Και αυτό καταδεικνύει ότι βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τη γεωρική ανάπτυξη. Και χρειαζόμαστε φυσικά ένα ολιστικό σύστημα για να υπάρξει ένα σύγχρονο, δυναμικό και ζωηρό περιβάλλον στην Ήπεθρο που να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία και να διασφαλιστεί έτσι το μέλλον και τη γεωργία και αυτών. Και γι' αυτό προτείνω πολλά στη μεταρρύθμιση του 2020. Η διατήρηση των φυσικών πόρων φυσικά θα βοηθήσει να έχουμε και ένα βιώσιμο μέλλον. Και στην κοινή γεωργική πολιτική, ο πρώτο τομέα περιβαλλοντική ε, ε σημαίνει ότι πρέπει να ε, ε, επενδύσουμε στο πρασίνισμα και στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους για να είναι πιο αποδοτικοί ενεργειακά. Και πολλές από τις ενέργειές μας έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές και τον εξχρονισμό. Και είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Έχουν μειωθεί κατά 20% εκπομπές αερίων ε, θερμοκηπίου από το 1990. Σε κάποιους ε, τομείς βέβαια μπορεί να αρχίζουν να ξανααυξάνονται. Αυτό μας ανησυχεί, διότι βελτιώνεται κατά πολύ η βιολογική γεωργία σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι 20% και ένα μεγάλο ποσοστό είναι αντικείμενο εκμετάλλευση ε, με βάση οικολογικά κριτήρια όπω η βοήθεια στη βιοπικιλότητα. Έχουμε ένα νέο κανονισμό για τη βιολογική γεωργία που θα αρχίσει να ισχύει το 2021 που θα εναρμονίσει του κανόνε και θα βοηθήσει του γεωργού με τα σύγχρονα μέσα που θα του βοηθήσουν να επεκταθούν περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία δεν είναι μόνο βιώσιμη, αλλά και ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. Το Δεκέμβριο του 2018 συμφωνήθηκε η οδηγία της Κομισιόν για τις ε, αθέμητες πρακτικές. Έτσι θα ενισχύσουμε τη θέση του Γεωργού στην τροφιμική αλυσίδα και θα βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας γενικότερα από την αθέμητη συμπεριφορά κάποιων που συμμετέχουν σε αυτήν την αλυσίδα. Οι Γεωργοί μας δίνουν ποιοτικά προϊόντα, αλλά και οι τιμέ του είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα με αυτά που λένε ορισμένοι, δεν φύγουμε την γεωργία στον αντισώμενο κόσμο. Υπάρχει ένα task force για τη γεωργία στην Αφρική, όπου αποδεικνύεται ότι κάνουμε βιώσιμες επενδύσεις και δημιουργούμε θέσεις εργασία στην Αφρική. Οι κύριοι εισαγωγοί των προϊόντων μα είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ελβετία. Ενώ εισάγουμε και πολλά προϊόντα. Είμαστε οι πρώτοι εισαγωγή από λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Τα περισσότερα μέτρα στήριξη τη κοινή γεωργική μα πολιτική δεν στρεβλώνουν το εμπόριο. Ούτω ή άλλω ε, είμαστε ο μεγαλύτερο εισαγωγέα γεωργικών προϊόντων από Αφρική. 3,6 δισεκατομμύρια εισήχθησαν από την Αφρική λοιπόν το 2018. Οι πολίτε μα δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την ασφάλεια των προμηθειών του ούτε να ανησυχούν για τη βιωσιμότητα. Και αυτό επίση συνδυάζεται με ένα λογικό και σωστό βιωτικό επίπεδο για του γεωργού μα. Η προσέγγιση μας λοιπόν για την κοινή γεωργική πολιτική λαμβάνει την υπόψη τη ε, αξιοπιστία, Διάβασα την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και αυτό επιβεβαιώνει ότι έχουμε μία όρημη και αποτελεσματική διαχειριστική δομή. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μετά το 2020 Θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω το αξιόπιστο σύστημά μα και προτείνουμε, όπω ξέρετε, μια νέα προσέγγιση. Όχι αυστηρού κανόνε συμμόρφωση, όχι αυστηρού γραφειοκρατικού κανόνε. Να περάσουμε σε αποτελέσματα και αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσά προσωπικά και τη Γενική Διεύθυνσή σας για το γεγονό ότι πάντοτε ε, mm. ανταποκρινόσασταν στα ερωτήματα της ε, Επιτροπή Κόντ αν και ως ε, εισηγήτρια ε, χρειάστηκε και θέλω και αυτή τη στιγμή να σας θέσω και κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Ακούγοντά σα, ε, ε, δημιουργεί, ε, σχηματίζει κανεί την εικόνα ότι όλοι οι γεωργοί μα θα έπρεπε να είναι κατενθουσιασμένοι. Ε, σας λέω όμως ανοιχτά ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Αντιθέτως, σε πάρα πολλά κράτη-μέλη συναντώ γεωργού οι οποίοι ε, λόγω του τεράστιου όγκου γραφειοκρατικών εργασιών που πολλές φορές είναι και αντιφατικές ε, ή έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Το ελεγκτικό συνέδριο τονίζει επανειλημμένος και δικαίως ότι θα πρέπει κανείς ε, να θεσπίζει οδηγίες και κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμοι Κατανοητή και να μην έρχονται αντίθεση ο ένας με τον άλλον. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε δυστυχώς ε, στον τομέα της γεωργίας. Ιδίω όσον αφορά το γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας. Από τα, από τα τελείως καθημερινά και πρακτικά πράγματα, τα, τις υποχρεώσεις που βαρύνουν έναν γεωργό έως και τα πιο σύνθετα, έως και τις πιο σύνθετες διαδικασίες, ε, όλα αυτά δημιουργούν ε, προβλήματα, γιατί ε, πολλές φορές δεν υπάρχει και διάκριση. Ε, το να, είναι σφάλμα το να μην έχει βάλει κανείς είναι ίδιο σφάλμα, ίδιο επίπεδο σφάλματος το να, βάλει κανείς τρεις μέρες ε, αργά την σήμανση στο αυτή ενό ζώου με το να μην το κάνει καθόλου. Αυτό καταλαβαίνετε ναι. ότι είναι μια τεράστια επιβάρυνση για τι ε, γεωργικές, τις αγροτικές οικογένειες και αυτό θα θέλαμε εμεί ω ε, Επιτροπή ε, Κοντ να απλουστευτούν οι διαδικασίε. Δεν μπορεί ένα γεωργός να πρέπει να έχει βγάλει πανεπιστήμιο για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Οπότε θέλω να σας ε, τονίσω και να σας καλέσω για άλλη μια φορά να προχωρήσετε σε αυτή την απλοποίηση εν ώψη του νέου πολίτες, δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, ε, διαπιστώσατε προβλήματα όσον αφορά την πιστοποίηση βιολογικών γεωργών. Ξέρετε ότι τα βιολογικά προϊόντα στην αγορά διατίθενται σε υψηλότερη τιμή και είναι και υψηλότερη η κερδοφορία που τα συνοδεύει. Όμως όταν υπάρχουν απάτες, τότε πρέπει κανείς να αναρωτηθεί ποιε είναι οι αιτίες ε, αυτών των περιπτώσεων απάτης. Πώς γίνεται, πώς λειτουργεί αυτή η απάτη, γιατί τελικά υπάρχει τέτοια κερδοφορία, γιατί παρακινείται κόσμος να προβεί σε απάτες. Τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν, τι πρέπει να κάνει η δική μας Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όταν θα έχει ένα προϊόν ένα σήμα βιολογικό, να είναι και πράγματι βιολογικό. Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε, τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν ε, οφείλονται σε αμέλεια, είναι απλά, αν θέλετε, σφάλματα ή αν πρόκειται για σοβαρές περιπτώσεις. Επίσης, στη Σλοβακία είχαμε περιπτώσεις που, και θα έλεγα το ίδιο και για τη Ρουμανία, πολλές φορές ε, με ευγενικό τρόπο, με εύσχυμο τρόπο αποκαλούνται ως double claims, διπλές αξιώσεις ότι πολλές φορές οι παρατυπίες αυτές δεν οφείλονται σε βούληση του ίδιου του γεωργού ότι πρόκειται για απλά σφάλματα ε, βλέπω ότι εδώ τα πράγματα βελτιώθηκαν από άποψη κομισιών και όσον αφορά τα κτηματολόγια Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν δυνατότητες για να ε, προβαίνει κανεί σε τέτοιε απάτη. και δυστυχώς ε, το κράτος δικαίου εδώ, σε αυτό το τομέα, δεν λειτουργεί με τον επιθυμητό τρόπο. Γι' αυτό και το ερώτημά μου προς εσά είναι πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι στη Σλοβακία, στη Ρουμανία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη θα σταματήσει η αρπαγή της γης και ότι εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις να επιβληθούν τόσο, σοβαρές, τόσο σοβαρά πρόστιμα ώστε κανείς πλέον να μην θεωρεί ότι ε, αυτό θα μπορούσε να είναι μια οδός κερδοφορία για τον ίδιο. Αποτρεπτικά δηλαδή. Δεύτερη παράκληση. Θα ήθελα, και χωρίς να θέλω να, να μου απαντήσετε σήμερα, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, όμως θα αποστείλω αυτό το ερώτημα και σε όλες τις γενικές διευθύνσεις. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε ε, συνολικά ε, πώς ε, υπολογίζεται το ποσοστό σφάλματος, με βάση ποιους ορισμούς, με βάση ποιους ελέγχους. Γιατί από γενική διεύθυνση σε γενική διεύθυνση ε, εμφανίζονται διαφορές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν διαβάζουμε ποσοστά σφάλματος, δεν γνωρίζουμε σε ποια βάση έχουν γίνει οι υποθέσεις αυτές, ποια δεδομένα έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταλήξει κανείς σε αυτά τα συμπέρασμα και πώς το συνολικό σύστημα ε, προσδιορισμού του ποσοστού σφάλματος τελικά είναι δομημένο. Νομίζω ότι είμαι σχετικά έξυπνη, αλλά πραγματικά με δυσκολεύει πάρα πάρα πολύ το να διαβάζω αυτά τα συστήματα των, του υπολογισμού των ποσοστών σφάλματος. Είναι δύσκολο καθήκον να, να, να, να, να το κάνει κανείς αυτό. Γι' αυτό και χωρίς να θέλω να μου απαντήσετε σήμερα, σας παρακαλώ κάποια στιγμή να μας αποστείλετε τις σχετικές πληροφορίες. Αυτά από εμένα. Βέβαια τα πλέον ενδιαφέροντα εσείς τα είπατε, οπότε ε, αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα στα οποία θέλαμε να, θα θέλαμε να μας απαντήσετε και από εκεί και πέρα θα ακούσουμε και άλλους ε, συναδέλφους που θέλουν να σας θέσουν ερωτήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αρχίζω λέγοντας ότι συμφωνώ μαζί σας. Όχι, δεν περιμένω τέτοια πράγματα από τους Γιώργους. Ποτέ δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Ποτέ δεν βρήκα έναν που να είναι ικανοποιημένο. Έτσι, αυτή είναι η φυσική του τάση. Πάντως, να σας απαντήσω στις ε, ερωτήσεις. Με 410 δις για επιταετία. εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Τέλος πάντων. γραφειοκρατία. Α, ακριβώς γι' αυτό κάνουμε τη μεταρρύθμιση. Από το 14 όπου πήγα μόλις είχαν νομοθετήσει μετά τη μεταρρύθμιση και ήδη είχαν αρχίσει τα παράπονα εγκρίνια για τη δυσκολία και για τη γραφειοκρατία. Ε, κανένας δεν συμφωνεί. Να φύγουμε από την προσέγγιση την νομοθετική ε, και να πάμε στην ε, προσέγγιση των επιδόσεων θέλουν όλα να τα κάνουν οι Βρυξέλλες. Γι' αυτό έκανε και αυτές τις προτάσεις. Αλλά πρέπει να θωρακίσουμε τον προϋπολογισμό, την πολιτική μας, την κοινή πολιτική. Αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να λάβουν τις ευθύνες τους οι περιφέρειες και τα κράτη. Εντάξει, τα βασικά εμείς τα αποφασίζουμε, αλλά τα επιμέρους τα κράτη-μέλη. Φαντάζομαι τα ξέρετε κι εσείς από τη Βαβαρία. Πριν από τρία χρόνια έλυσε ένα πρόβλημα που υπήρχε και δόθηκε τότε ο ορισμός του ανθρωπίνου σφάλματος και ανατομία στο, στη, νομική επιστήμη. Και έτσι προχωρήσαμε και έλυσε... Α, πολύ χαίρομαι που ξέρετε τα της Βαβαρίας. Ε, βέβαια τα ξέρω αυτά που έχω λύσει. Όπου έδωσα λύση τα ξέρω τα προκέτσι και έκανα 150 αλλαγές και απλουστεύσεις από το 14 και οι προτάση για το 20 είναι να μειωθούν κάποια μέτρα από 17 σε 8 και από 200 τόσα να πάνε σε λιγότερα από 50 όσον αφορά την κοινή αγορά. Την κοινή οργάνωση αγοράς τέλος πάντων. Και να φύγουμε από αυτήν την εφαρμογή της προσήλωσης στον νόμο ε, που φοβίζει τόσο πολύ τα κράτη-μέλη γιατί θα πρέπει όλα να γίνουν όπως πρέπει και ένα σωρό μέτρα για τον προπολογισμό, αλλά τότε τα μικρά σφάλματα είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί υπάρχει απώλεια εισοδήματο από τι εκμεταλλεύσει. Αλλά αν πάμε προ τα εκεί, τότε μειώνουμε το πρόβλημα και θωρακίζουμε τον προπολογισμό. Βιολογικέ καλλιέργειε, ακριβώ λόγω τη απάτη, αλλάξαμε τον οργανισμό που αρχίζει από το 21, σημαντικό νομοθέτημα. Ο Μάρτιν Χάσινγκ ήταν ο εισηγητής νομίζω είναι σωστή συμφωνία, να υπάρχει ισονομία, ε, δίκαιοι κανόνες, οι εισαγωγέ και και μετά είχαμε εκτό από τη Γερμανία πρόβλημα και με τις κάτω πάτες πάτε, όλα αυτά τα εφαρμόσαμε και οι έλεγχοι εφαρμόστηκαν από τα κράτη-μέλη και τα πράγματα βελτιώθηκαν. Γενικά, οργάνωση των ελέγχων γίνεται από τα κράτη-μέλη και έτσι να είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους Γιώργους. Νέο σύστημα προληπτικών ελέγχων. Και τώρα μπορούμε ιντερνετικά να ελέγχουμε. 6.000 ήταν οι Γιώργοι που ωφελήθηκαν, αλλιώς θα είχαν πέσει σε κάποια λάσσονα σφάλματα και θα είχαν πληρώσει πρόστιμα. Άρα, το θέμα δεν είναι να κυνηγήσουμε τον κόσμο, αλλά να τους δώσουμε κίνητρο συμμόρφωσης. Γιατί να πάτε τώρα, για τις σημαντικές περιπτώσεις είναι άλλος τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι η διασταυρούμενη συμμόρφωση και οι εθνικοί κανόνες εν προκειμένου. Και όλα πηγάζουν από την ε, νομοθεσία της ΚΑΠ. ξέρω ότι σας απασχολεί ο αριθμός των ελέγχων, ε, περισσότερα έλεγχοι στην ίδια εκμετάλλευση. 5% των ελέγχων έχουμε τώρα, οπότε και έχουμε μεγάλο ποσοστό σφάλματος και εκεί ε, βλέπουμε ε, να υπάρχει μια τάση μη συμμόρφωσης και ελπίζουμε θα πέσουμε 1% αλλά άρα και επιδόσεις έχουμε και αποτελέσματα. Και έτσι προσπαθούμε να κάνουμε και τη διοίκηση και, τους, και τις εκμεταλλεύσεις να είναι σωστοί. Έξι κρατημέλη μείωσαν τους ελέγχους και άλλο ένα κράτος μέλος. Ε, προσχώρησε σε αυτή την τάση το 19. Η τελική ευθύνη και η τελική απόφαση λοιπόν θα είναι κάτι που θα απόκειται στα κράτη-μέλη. Σλοβακία και Ρουμανία. Ισχυρισμοί, καταγγελίες για ε, απάτες. Έρευνα από την Όλαφ. Και έγινε η διαφοροποίηση από την Όλαφ και να ξέρει ο κόσμος ότι αν έχουμε ελέγχους διαχείριση είναι η Άγκρη, είναι απάτη η Όλαφ και οπότε έχουμε ένα πρόγραμμα για την ε, Σλοβακία. Συνεχίζονται οι οικονομικοί έλεγχοι. Τώρα στη Σλοβακία θα γίνουν διορθώσεις όσον αφορά τον οικονομικό κίνδυνο για την Ένωση. Και έχουμε την κατά την παράσταση ε, διαδικασία και οι αρχές μπορούν να επιχειρηματολογήσουν για ό,τι βρήκαμε και προσπαθούμε όπου καταλήξουμε αυτό να είναι κάτι που να στέκει στο δικαστήριο. Άρα πολύ σοβαρά βλέπουμε αυτή την υπόθεση γιατί είναι σοβαρή. Και ο... η διευθύντρια εδώ είναι εκ δεξιών μου και έχει έρθει εδώ την ξέρετε αλλά έχει πάει προσωπικά στους κονικούς ελέγχους στη Σλοβακία ούτως ώστε να φέρουμε εις πέρα στη διαδικασία σωστά στη Ρουμανία τώρα. Στην αρχή μετά την ε, προσχώρηση τα πράγματα ήταν δύσκολα για τη Ρουμανία, τώρα όμω έχουν μεγάλη απορρόφηση των άμεσων πληρωμών, 98,8% το 18-99% φέτος πάνω από τον μεσόρο 53% Το θέμα είναι αυτό, η φαρπαγή της γης σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη Ξέρετε τι γίνεται στην Σλοβακία. Αλλά έχουμε αναλάβει δράση και εκεί. Αλλά όταν έχουμε ισχυρισμούς για παράνομες πρακτικές, ψάχνουμε και καμιά φορά πιστεύουμε δεν γίνεται τίποτα. Άλλοτε όμως βρίσκουμε. Οπότε όταν μια διαδικασία συνεχίζεται την αφήνουμε να ολοκληρωθεί. Τώρα για την υφαρπαγή της γης. Έχουμε 8% στη Ρουμανία της γης. Μεγάλες εκμεταλλεύσεις. 3 εκατομμύρια γεωργία. Κάτω από τα 5 εκτάρια. Οπότε όταν έχουμε τέτοιου ισχυρισμού για αρπαγή τη γη, ε, τότε είναι θέμα κράτου μέλου. Αλλά εμεί τώρα δούμε τι γίνεται με τι πληρωμέ, που είναι άλλο θέμα, αν υπάρχει και απάτη. Βλέπουμε το σύστημα διαχείριση ελέγχου. Και γνωρίζω μια περίπτωση, μια υπόθεση κάποιο κράτο μέλο που υπήρχε ανησυχία για αρπαγή της γης. Αλλά πρέπει να υπάρχουν καταγγελίες και αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Καταγγελίες και στοιχεία. Διαβάζουμε στα ΜΜΕ, ε, αλλά χρειάζεται η καταγγελία του. Οπότε για το ποσοστό σφάλματος. Αν κάτι δεν σας αρέσει όταν συγκρίνετε συμπεράσματα γενικών διευθύνσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Διευθύντρια και θα το υπολογίσουμε. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το... Λοιπόν, Ισκιώδη. Πρώτα απ' όλα, συνάδελφος Πένκοβα, σοσιαλίστρια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε Χόγκαν. Πάρα πολύ πλήρης οι απαντήσεις σας. Για να δούμε τώρα κάποια θέματα για το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις σας. Πρώτα-πρώτα. Οι επιλογές ή απλουστευμένες για το κόστος της δαπάνης και την ΚΑΠ. Τα κράτη-μέλη έχουν θέματα για την υλοποίηση του μέτρου. Έχουμε ένα σωρό ενέργειες της Κομισιόν για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτή τη διαδικασία και τις κατευθυντήριες που έχετε εξαγγείλει για αυτή την ε, περίοδο προγραμματισμού. Αλλά για την επομένη δεν λέτε το αν υπάρχουν τέτοιες κατευθυντήριες και σε σχέση με το τι ζητούν τα κράτη-μέλη θα γίνουν ε, αλλαγές. στο Γιατί δεν έχετε δώσει καθεντήριες για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Δεν φοβάστε ότι έτσι θα επιβραδυνθεί η διαδικασία και πάμε για περισσότερα λάθη. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη, σύντομη. Για την επιστροφή τη βάση των αποτελεσμάτων δύναμη του κανονισμού του 18 που επιτρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση που να μην συνδέεται με τις δαπάνες αλλά συνδέεται με την συμμόρφωση, με τις επιδόσεις και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θέλει να γίνει μια κατεξοδότηση πράξη όσον αφορά το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης πέραν των αρχικών ε, πόρων των Ταμείων Ανάπτυξης. Όμως στην απάντησή σας λέτε ότι μετά αξιολόγηση δεν θα εφαρμόσετε την κατεξοδότηση πράξη για το Ταμείο Ανάπτυξη της Υπέθρου. Όμως επίσης μας λέτε ότι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να έχουν ε, μια προσέγγιση σε σχέση με την επίτευξη των επιδόσεων. Για τα άλλα ταμεία, τους άλλους πόρους τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη. Πώς στην πράξη όλα αυτά θα υλοποιηθούν, πώς θα βοηθήσετε. Θα συνεργαστείτε με το ελεγκτικό συνέδριο για αυτό το ζήτημα. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολιβιέ Σαστέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ προφανώς να σας ευχαριστήσω για την ε, συμμετοχή σας εδώ και για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης δραστηριοτήτων ε, της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη. Είναι σημαντική για μας. Είναι συνέχεια της ενημέρωσης που μας έκανε το ελεγκτικό συνέδριο για ορισμένα στοιχεία του 2018. Δεν, δεν θα υπενθυμίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η Γενική Διεύθυνση από πολλέ απόψει. Ε, πρώτα απ' όλα έχει σημαντικό προπολογισμό και είναι πολύ σημαντική βέβαια και η κοινή γεωργική πολιτική για το μέλλον των γεωργών και φυσικά και η ανάγκη οι καταναλωτέ στην Ευρώπη να έχουν ε, ποιοτικά προϊόντα, διαφορετικά προϊόντα, σε λογικέ τιμέ. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι διαχειρίζεστε 59 δι, 37% του προπολογισμού του 2018. Η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, όπω ακούσαμε, λέει ότι το ποσοστό σφαλμάτων είναι 2,4% για του φυσικού πόρου το 2018. Ναι, βεβαίω. Το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των προηγουμένων ετών. Αλλά είναι αξιόλογο. Και στις άμεσες πληρωμέ δεν έχουμε βέβαια τόσο, σημαντικές, ε, τόσο σημαντικά σφάλματα με βάση τις, ε, τους ελέγχους του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά η περιπλοκότητα των ευρωπαϊκών κανόνων και η περιπλοκότητα των κανόνων των κρατών μελών αυξάνει τον κίνδυνο σφαλμάτων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει. Όσο πιο περίπλοκοι είναι οι κανόνες, τόσο διαφορετικότερες είναι οι ερμηνείες τους και άρα υπόκεινται περισσότερο σε σφάλματα. Και ξέρουμε ότι 99% του υπερπολογισμού είναι κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Οπότε η προσπάθεια απλούστευσης πρέπει να είναι μόνιμο μέλημα, διότι Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και να απλουστεύσουμε και να μειώσουμε και τα σφάλματα. Τώρα, να κάνω μερικές συγκεκριμένες ερωτήσει. Διαβάζω ότι το ηλεκτρικό συνέδριο μας είπε ότι υπήρξαν απτές ανεπάρκειες στις εργασίες των ε, οργανισμών, των φορέων πιστοποίησης. Θέλω τη γνώμη σας για αυτό το θέμα. Το συνέδριο πάντα επανειλημμένα τονίζει ότι οι δείκτε αποτελεσμάτων δεν είναι πάντα οι πιο κατάλληλοι για την ανάπτυξη τη υπαίθρου, τους νέου γεωργού τις πληρωμές. Δεν έχουμε επαρκείς ε, δείκτε και για το πρασίνισμα. Τώρα που ολοκληρώνεται η θητεία, τι κάναμε τα τελευταία χρόνια. Και για το μέλλον, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τη μέτρηση των αποτελεσμάτων, της ε, αποτελεσματικότητα των αποτελεσμάτων. Τώρα, ετήσια έκθεση δράση. Μα εξηγείται ότι ορισμένες συστάσεις των εσωτερικών ελέγχων πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν. Εγώ θα προτιμούσα να μας πείτε γιατί δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Ήδη εξηγήσατε, απαντώντας σε ερωτήσεις ε, συναδέλφων, εκφράσατε τη βούλησή σας να απλουστεύσετε τους διοικητικούς κανόνες, δεν θα επανέλθω, αλλά η καταπολέμηση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο στη Γεωργία. Ναι, ελήφθησαν κάποια μέτρα. Αλλά πάντα στην ετήσια έκθεση λέγεται ότι οι εκπομπέ διοξιδίου αυξήθηκαν μεταξύ του 2015 και του 2016. Ενώ για το 17 και το 2018 δεν έχουμε στοιχεία. Μήπω τα έχετε εσεί, μήπω μπορείτε να μα τα δώσετε. Πώ είναι δυνατόν να αυξάνονται οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα μεταξύ 15 και 16. Επίσης, ποια είναι η αξιολόγησή σας για τα λεγόμενα EU Action for Smart Villages, για τα ευφυή e χωριά, για να υπάρξει περισσότερη ψηφιοποίηση της γεωργίας. Γιατί συνδέεται με τις ερωτήσεις μου. Διότι οι διαδικασίες πληρωμών μέσω του ίντερνετ προφανώς μειώνουν ε, το ενδεχόμενο σφάλματος πώς θα διευρύνετε και θα κατοχυρώσετε αυτή τη μέθοδο πληρωμών που σίγουρα θα βοηθούσε και σε απλούστευση και σε μείωση των σφαλμάτων. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Πίτροπε, θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, γιατί άμα γίνουν πάρα πολλές, Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για τις ε, απλοποιημένες ε, ενελακτικές δυνατότητες κόστου. κόστους. Το συνέδριο λέει ότι έτσι μειώνει γραφειοκρατία. Άρα οι απλουστευμένες επιλογές κόστους είναι καλύτερες. Και τονίζω ότι αυτές οι απλουστευμένες ε, επιλογές κόστους επιτρέπουν ταχύτερα να καθοριστεί το ύψος ε, των επιστροφών και άρα μας επιτρέπουν να εστιάσουμε περισσότερο στην εφαρμογή της πολιτικής. Το κάναμε και μέσω του κανονισμού Omnibus πριν από δύο χρόνια εν μέρη. Και έτσι τα κράτη-μέλη έχουν περισσότερη αυτονομία και περισσότερες πιθανότητες να αξιοποιήσουν αυτές τις απλουστευμένες επιλογές. Τώρα για την ε, επαλήθευση της μεθοδολογίας και για τον υπολογισμό αυτών των απλουστευμένων εναλλακτικών. Βεβαίω, ε, οι οργανισμοί πιστοποίηση δίνουν ήδη γνώμη, γνώμη για την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών και την εφαρμογή του νόμου για αυτέ τι απλουστευμένε επιλογέ κόστου. Όλε οι συστάσει λοιπόν έχουν γίνει δεκτέ. Και οι δράσει είναι ήδη σε φάση εφαρμογή ή ε, ολοκληρώνεται η εφαρμογή τους. Τώρα, για την ε, κατεξοδότηση πράξη. Είναι η DG Regi αρμόδια, αλλά εμείς τους δίνουμε βοήθεια. Και συνεργαζόμεθα ήδη και με το ελεκτικό συνέδριο για τις ειδικέ εκθέσεις και για καταλόγους με το τι πρέπει να γίνει, checklist. Συνεργαζόμεθα λοιπόν με την DG Regio. Τώρα, δεν είναι σωστό να έχετε την εντύπωση ότι δεν θα δίνουμε τεχνική βοήθεια για τη νέα μεταρρύθμιση. Μα θα, θα δίνουμε, θα δώσουμε. Και ήδη δίνουμε. Ω DG Agri σε όλα τα κράτη-μέλη. Με διάφορου τρόπου. Έγραφα με καθευτήριε γραμμέ, ε, σεμινάρια. Προσπαθούμε να του βοηθήσουμε να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να υιοθετήσουν τις στρατηγικές τους για την κοινή γεωργική πολιτική με τον νέο τρόπο εφαρμογής. Βεβαίω. όσο πιο περίπλοκα είναι τα συστήματα, τόσο περισσότερο θα είναι τα σφάλματα. Αλλά εάν περάσουμε σε μέτρηση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης, τότε θα μειωθούν πολύ τα μικρά λάθη και θα είναι πιο στόχο προσιλωμένη η προσέγγιση μας. Τώρα, η εσωτερική έλεγχοι. Πώς λειτουργούν, με ρωτήσατε. Έχουμε εσωτερικούς ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα σύστημα. Ελέγχει περιοδικά την εργασία των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Και μέχρι τον ε, επόμενο Δεκέμβριο πρέπει να εφαρμόσουμε έξι συστάσεις τις οποίες εφαρμόζουμε με βάση τα σχέδια δράσης που έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη. Άρα δεν, είναι, δεν εκκρεμούν αυτές οι συστάσεις. Είναι σε διαδικασία εφαρμογής. Όλα όσα λένε τα σχέδια δράσης τα εφαρμόζουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Σαστέλ ότι είναι περίπλοκη πολιτική. Το είπα στις απαντήσεις μου στην Πρόεδρο. Οι φορείς ε, πιστοποίησης κάνουν τη δουλειά τους και έχουμε σημειώσει πρόοδο προς την προσέγγιση ενιαίου ελέγχου. Έχουν υπάρξει τέσσερις περίοδοι εφαρμογής αυτής της διαδικασίας και πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί η αξιοπιστία. Για το οικονομικό έτος 2018 οι φορείς αξιοπιστίας έδωσαν περισσότερη συμβολή στην προσαρμογή του ποσοστού στην προσαρμογή του ποσοστού σφαλμάτων. Κοιτάξτε, έχουμε σχέδια δράσης. Οι έλεγχοι του συνεδρίου των κρατών μελών μπορεί να μην βρουν λάθη. Αλλά εμεί λαμβάνουμε υπόψη αυτά που βρίσκουν και οι οργανισμοί πληρωμών. Όλοι λοιπόν συνεργαζόμεθα. Άρα, ό,τι ξεφύγει από τον ένα το πιάνει ο άλλο. Συλλογικά. Και βλέπουμε και τι βελτιώσει πρέπει να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να βοηθούμε τους ε, φορείς πιστοποίησης. Αυτή η μεταφορά του κέντρου βάρους στην ε, απόδοση και τα αποτελέσματα δεν είναι καινούργια. Το κάνουμε ήδη για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου. Κάποιοι πόροι που θα στείλουμε στα κράτη-μέλη θα σταλούν για καλή απόδοση των προγραμμάτων του πυλώνα 2. Και θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την προσέγγιση και στον πυλώνα 1. Γιατί υπάρχουν τόσοι και οριζόντιοι στόχοι που εξαρτώνται από την αιρεσιμότητα. Και θα έχουμε και δείκτες που θα μας δείχνουν αν λειτουργεί το σύστημα. Και θα θέσουμε και στόχους και ορόσημα. Τα κάνουμε ήδη στην περιβαλλοντική πολιτική. Οι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα. Είπε ότι υπήρξε μείωση 20% από το 1990. Συμφωνώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Υπήρξε σε ορισμένου τομεί αντιστροφή αυτή τη θετική πορεία. Θα το αντιμετωπίσουμε. Και ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία υπάρχουν προβλήματα. Τα ευφυή χωριά είναι κάτι που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Και μέσω τη δήλωση για την ανάπτυξη πέθρου, ο κύριος Μπόκοβιτς και ο πρώην Ευρωβουλευτής Τσάνι έκαναν πολύ καλή δουλειά, λειτουργήσαν πιλωτικά προγράμματα για τα ευφυή χωριά. Αυτό μας κάνει να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η συνδεσιμότητα και ιδιαίτερα η ευρυζωνικότητα. Είπα ότι έχει ανέβει στο 53% στην Ήπεθρο, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και τελευταία ερώτηση. Χρήση τεχνολογίες για να γίνονται επιγραμμικά οι αιτήσει. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2020 να έχουμε 100% ηλεκτρονικές αιτήσει παντού, σε όλα τα κράτη-μέλη. θα βοηθήσει τους γεωργούς θα μειώσει την ε, περιπλοκότητα, θα μειώσει τα μικρή κλίμακα σφάλματα. Μέχρι τέλου του 2020. Κάποια κράτη-μέλη, εντάξει, θέλουν κάποια παράταση για να αρχίσουν να λειτουργούν τα συστήματά τους, αλλά ελπίζουμε μέχρι το 2021 να το έχουν επιτύχει όλοι. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Όλα των κράμων είναι η επόμενη Ισκιώδης. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, καλύτερα να μιλήσω γερμανικά για να είμαι και λίγο πιο ακριβής σε αυτά που θέλω να πω. Λοιπόν, είπατε μόλι ότι υπάρχουν δείκτες ε, στον ε, τομέα του περιβάλλοντος που θέλετε να εφαρμόσετε και στις μεταρρυθμίσεις κοινή γεωργικής πολιτικής. Υπάρχουν όμως ήδη κάποιες μορφές δικτών για την αξιολόγηση και, τον, και της τρέχουσας κοινή γεωργικής πολιτικής. Και όχι μόνο το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και πολλά, πολλοί επιστημονικοί φορείς τον τελευταίο καιρό Ε, έκαναν μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρασινίσματος. Και τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που μας παρουσιάσατε εσείς. Ήταν πραγματικά εξοντοτικά ε, τα, τα αποτελέσματα αυτά. Και θέλω πραγματικά να επικεντρωθώ σε αυτό. Το πρασίνισμα της του πρώτου πυλώνα. 73% του γεωργικού προπολογισμού ακόμη κατευθύνονται στον πρώτο πυλώνα. Μιλάμε δηλαδή για 30,5% του συνολικού ενωσιακού προπολογισμού, ο οποίος ε, κατευθύνεται στον πρώτο πυλώνα και αναρωτιόμαστε αν το πρασίνισμα είναι κατά 90% αναποτελεσματικό, γιατί τότε δεν επιδιώκουμε μια θεμελιώδη μεταρρύθμιση του πρώτου πυλώνα. Γιατί υποβάλλει η Κομισιόν πρόταση μεταρρύθμισης που προβλέπει μείωση του πρώτου πυλώνα κατά 11% αλλά εκεί όπου πραγματικά είναι αποτελεσματικά τα πράγματα, εκεί που υπάρχουν περιβαλλοντικά μέτρα εκεί που πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε αποτελεσματικά περιβαλλοντικά μέτρα στο δεύτερο πυλώνα εκεί προτείνεται, 28% μείωση. Αυτό ούτε εμπειρικά ούτε επιστημονικά μπορεί κανείς να το θεμελιώσει. Ε, αν δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ε, στα σοβαρά και τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, ε, θα, δούμε ότι έρχονται σε αντίθεση αυτά που προτείνεται ακόμη και με τη συνθήκη. Πώς λοιπόν οι προτάσεις σας κινούνται σε απολύτως αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της αποτελεσματικότητας. Αυτό το είδαμε και με τα συστήματα ECOS. Όταν χρειάζεται η, η σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών, τότε πάντοτε θα έχουμε να κάνουμε με τον ελάχιστο κοινό παραμε παρονομαστή. Και αυτός ο ελάχιστος ε... Ε... κοινός παρονομαστής δεν ενισχύει ούτε τις επιδόσεις, ούτε την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, ούτε την προστασία της ευδοίας... ευζοίας των ζώων, ούτε την ε, προστασία του κλίματος. Γι' αυτό και έχω πολύ μεγάλες ε, διαφωνίες σε σχέση με τα όσα μας είπατε εσείς και περιγράφοντας την τελευταία επταετία. Δεύτερον, ομολογώ ότι μου φάνηκε αρκετά κοινικός ο τρόπος που απαντήσατε για τη, στην ερώτηση της Προέδρου για τη Σλοβακία και τη Ρουμανία. Μας είπατε ότι δεν λάβατε καταγγελίες ή παράπονα από τους γεωργούς. Μα ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η δομή της γεωργίας στη Ρουμανία. Είπατε εσείς ο ίδιος ότι υπάρχουν μόλις 8% μεγάλες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι άνω των 90% ε, όμως των επιχορηγήσεων στον αγροτικό τομέα κατευθύνονται σε αυτές τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις. 600.000 ε, αγρότες στην Ρουμανία λαμβάνουν 46 ευρώ το χρόνο. Τι σημαίνει αυτό, ότι το μεγάλο, το, η μερίδα του λέοντος των γεωργικών ενισχύσεων πηγαίνουν σε 8, 10, 20 ε, μεγαλοκαρχαρίες σε, δικαιού, σε δικαιούχους μεγάλους. Αυτό τι σημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν επιτρέπει στους μικρούς γεωργούς να απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Μα δεν έχουν καν τη δυνατότητα. Ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Πηγαίνουν οι, οι ολιγάρχες ε, της γης και εκβιάζουν, αρπάζουν τη γη από τους μικρούς γεωργούς. Δική σας δουλειά ως Επιτρόπου θα ήταν να δημιουργήσετε μια υπηρεσία όπου θα μπορούσαν να ε, τίθενται σε επεξεργασία τέτοια, τέτοια παράπονα, τέτοιες καταγγελίες. Λέτε ότι δεν λάβατε καταγγελίε. Μα φυσικά και δεν λάβατε, αφού δεν έχετε προβλέψει δομέ για την παραλαβή τέτοιων καταγγελιών. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα της κατανομής των κονδυλίων. Πρόεδρος, να συμπληρώσω κι εγώ, γιατί έχω πάει κι εγώ πολλές φορές στη Ρουμανία. Επίτροπε, είπατε βεβαίως ότι με βάση την αρχή της επικορικότητας ε, υπάρχουν εθνικές αρμοδιότητες κτλ. Ε, βέβαια είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όταν μιλάμε για τη Βαβαρία και την Ιρλανδία ή όταν μιλάμε για κράτη-μέλη στα οποία πραγματικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες. Όμως το να θεωρεί κανείς δεδομένο ότι το κράτος δικαίου στη Βουλγαρία, στη Σλοβακία και στη Ρουμανία ε, προστατεύει τους ε, γεωργούς ε, είναι σχεδόν ηρωνία. Χρειαζόμαστε βοήθεια στους γεωργούς και δεν κατηγορώ μόνο την, την Κομισιόν. Ξέρω ότι δεν θα μπορούσε η Κομισιόν να υποκαταστήσει όλες τις εθνικές αρχές που θα έπρεπε να επιτελούν αυτό το, το έργο. Το ερώτημά, μας, το ερώτημά μας όμως είναι τι αλλαγές πρέπει να γίνουν ώστε οι γεωργοί να λαμβάνουν τις αναγκαίες ε, επιχορογήσεις που δικαιούνται. Και πώς μπορεί η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να βασίζεται στο έργο των ε, φορέων πιστοποίησης. Ε, είπατε βεβαίως ότι μόνο το 25% αυτών των φορέων πιστοποίησης διαπιστώθηκε ότι είναι, άξιοπιστοί. είναι αξιόπιστη. Στα 20 μέτρα που προτείνεται για τη βελτίωση της κατάστασης μπορείτε να, μας, μπορείτε να μας τα περιγράψετε για άλλη μια φορά για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε και εμεί μια εικόνα ε, για το ποια είναι τα προβλήματα γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Κύριο Σιγόφσκι. I'm sorry, Συμπαθάτε με, αλλά ήμουν τόσο απροθυμένος από τις ομιλίες μας που ξέχασα ότι και εγώ θα πρέπει να σας πω τα δικά μου. Πρώτα πρώτα επίτροπε. Πρώτη φορά συμφωνώ μαζί σας. Να το γιορτάσουμε και ήταν τρομερή η ομιλία σας και βέβαια δυστυχώς εδώ είστε για τελευταία φορά αλλά αν κουβεντιάσουμε για την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτή την τελευταία σας εμφάνιση εδώ. Και αν ξανάρθετε θα είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Τώρα για το ερωτηματολόγιο. Πραγματικά για πρώτη φορά μπορώ να πω ότι οι απαντήσεις επιτρόπου στις συγκεκριμένες μας ερωτήσεις είναι συγκεκριμένες ως απαντήσεις και μπράβο, μπράβο σε εσάς και στο επιτελείο σας και δεν το λέω ειρωνικά. Το εννοώ είναι υπέροχο το ότι κανείς μπορεί να διαβάσει συγκεκριμένη απάντηση για τις ερωτήσεις μου το 3 ή το 4. Αλλά βέβαια θα μπορούσα να ρωτήσω και ακόμα πιο συγκεκριμένα από όσο μας εκτυπεί στην απάντηση και ρωτώ πότε θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, πότε θα έχετε κλειδώσει το θέμα του 18 για την ερώτηση παρθμών 4 Μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για τη νέα μεθοδολογία που μετέρχεται η ΑΠΑ. Είμαι πάρα πολύ σημαντικό να μάθω πώς το σκέφτεστε όσον αφορά επιπλέον κριτήρια για βιώσιμη και βιολογική γεωργία, φιλική προς το περιβάλλον. Βελτίωση όσον αφορά την διανομή και όσον αφορά την στόχευση των μεσών πληρωμών και πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση, χορήγηση πόρων, για ε, ε, χώρους στάθμευσης και σε σχέση με τη Γεωργία γιατί έχω κατά νου την υπόθεση της Σλοβακίας, αυτό που περνάμε τώρα και είδαμε στην επίσκεψη την αποστολή τέλο πάντων, άλλα θέματα Πόσες εκδηλώσεις ε, συνολικά οργανώσατε για νέου Γεωργού και πόσοι εξ αυτών συμμετέσχουν. Πολύ σημαντικά θέματα αυτά για μένα. Γιατί αφορούν πάρα πολλούς. Πάρα πολλοί δήλωσαν νέοι αγρότες και ξέρουμε τι γίνεται. Τα κριτήρια επιλογής τώρα είναι θέμα εθνικό, αλλά εσείς πώς εξασφαλίζετε το ότι οι πόροι όντως απορροφούνται, αξιοποιούνται από και για τους νέους ε, οργίους και όχι από άλλους. Ξέρω εγώ από συγγενείς τους. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Die Kollegin Rivasi wäre, würde den Abschluss... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Φιλ Χόγκεν, είστε αισιόδοξο μέσα σε μια δραματική κατάσταση πρώτα-πρώτα. Είστε ο πρώτο που εσεί ο ίδιο αναγνωρίζετε ότι είναι πολύ άνηση αυτή η ΚΑΠ. Γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για τι ενισχύσει σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό των μικρών γεωργών η ενδείξει για τον πρώτο και για το. Τα κριτήρια τα πούμε, για πρώτο και δεύτερο πυλώνα δεν λειτουργούν. Και τώρα κάτι άλλο, κύριε Φιλ Χόγκαν. Ντρέπαμε για το ότι αυτοκτονεί κάθε δύο μέρες ένας γεωργό. Επί δική σα θητεία ως Επιτρόπου Γεωργία. Ήσασταν, ήσασταν. Δεν περιφερόμαστε καθόλου αυτόν τον απολογισμό. Μας λέτε για τις επιχειρήσεις, μας λέτε διάφορα αλλά τίποτα για τους μικροκαλλιεργητές οι οποίοι ε, δεν συμμορφώνονται μετά του τους. Και υπάρχει ε, αυτού του είδους το βρέχει κύκλωμα στην παραγωγή. Άρα δεν τα πάτε και τόσο καλά. Για πέστε μου. Όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις και έχουμε 86% των Ευρωπαίων που θέλουν υγιή προϊόντα, δεν θέλουν λιπάσματα, θέλουν αντιβιωτικά, δεν θέλουν τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και αν ρίξει κανείς μια ματιά στο ενέκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μας τα είπε για τα βιολογικά προϊόντα η πρόεδρος και είναι ένα σωρό τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα αλλά τι γίνεται με τους παραγωγούς, πού είναι. Έχουμε 13% των ε, εισηγμένων, αλλά σε... πώς αντιστοιχούν σε κάποιους ε, στοχευμένους παραγωγούς. Αυτό έχει να κάνει με την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων, των βιολογικών. Τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο των ε, εισαγωμένων προϊόντων, ένα σωρό λοιπάσματα έχουν απαγορευτεί, αλλά παρόλα αυτά αυτά τα φυτοφάρμακα τα πουλάμε στην Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στη Βραζιλία και τι γίνεται στα πλαίσια των συμφωνιών. Ε, δίνουμε κάποια εκατότατα όρια ε, ανοχής, ανώτατα όρια ανοχής, αλλά ποιον δεν θα έπρεπε να είναι μηδέν, αφού τα έχουμε απαγορεύσει αυτά στην, ε, στις ουσίες πάντων στην Ευρώπη. Ένα αυτό. ότι υπάρχει επαρκής έλεγχος από πλευράς των ε, εισαγωμένων πλευρά των ε, κρατών μελών και το ίδιο ισχύει και για τα πρόσθετα στα είδη διατροφή. για τα βαρέα μέταλλα, του ενδοκρινούς διαταράκτες και το ίδιο ισχύει και για τις συσκευασίε και μας λέει το ελληνικό συνέδριο τι γίνεται. Έχουμε αναβάθμιση τη νομοθεσία επ' αυτών. Πώς έχουν τα πράγματα. Και το τελευταίο που μας λέει το ελληνικό συνέδριο είναι όσον αφορά την ΕΦΣΑ, την κοινοτική υπηρεσία λέει ότι δεν υπάρχουν τα μέσα ούτως ώστε να γίνουν κάποιες επιστημονικές έρευνες όσον αφορά τα κατάλοιπα των ε, φυτοφαρμάκων. Τι λέτε, τι προτείνετε. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρέπει να βρεθώ κάπως στον Επίτροπο, διότι του κάνετε ερωτήσεις που δεν είναι στο πεδίο αρμοδιοτήτων του. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα απαντήσει. Κύριε Επίτροπε, Άλλη επιτροπή είναι για τα ορισμένα από τα θέματα που θέσατε. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Μα εξεπλάγει που ο φίλος από ή φίλοι από το κόμμα των Πρασίνων επιτίθεται στην κοινή γεωργική πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει να εκπλήσουμε, γιατί ό,τι και να προτείνουμε, οι πράσινοι ποτέ δεν μα στήριξαν. Στην μεταρρύθμιση του 2013, που ήταν 30% για το πρασίνισμα, ήσασταν κατά, το καταψηφίσατε. Μα απαντάω στους ερωτήσει σα, κυρία μου. Είπατε πολλούς τομείς Αναφερθήκατε σε πολλούς τομείς όπου ε, έχουμε οικονομικούς και οικολογικούς στόχους ε, συμπεριλαμβανομένης της βιοπικιλότητας, ε, της υγιούς διατροφής, των σωστών περιβαλλοντικών πρακτικών. Αλλάζουμε την κατάσταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι λειτουργούν σωστά τα μέτρα πρασινίσματος, ούτε ότι είναι παρκώς φιλόδοξα. Και αν δείτε τις τωρινές προτάσεις, που δεν φαίνεται να τις έχετε διαβάσει, η αιρεσιμότητα στον πυλώνα 1 θα ισχύσει πολύ την ευθύνη των γεωργών για την εφαρμογή των μέτρων παρασυνίσματος. Ο συνολικός προβλημό της ε, κοινή πολιτικής θα πρέπει να ασχολείται με τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Θα έχουμε εκο-προγράμματα για τα προγράμματα δράσης των κρατών μελών με βάση αυτά που προτείνετε κι εσείς. Στον πυλώνα 1 θα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για οικολογικά προγράμματα και στον πυλώνα 2 στηρίζετε τα μέτρα για το περιβάλλον. Εδώ όμως ε, και εμείς έχουμε βελτιώσει τους ε, στόχους, αυξήσει τους στόχους, εξαιρώντας κάποιες περιοχές που έχουν ε, ειδικά προβλήματα. Υπάρχει τεράστια αύξηση λοιπόν στην φιλοδοξία της προσέγγισής μας για το περιβάλλον. Και τα στοιχεία που δίνεται είναι λάθος για αυτά που λέμε στον προπολισμό. Τα στοιχεία είναι 4,6% για τις πληρωμές του πυλώνα 1, σε τρέχουσες τιμέ. Εσείς αναφερθήκατε σε τιμέ ε, προσαρμοσμένες ε, στον πληθωρισμό, αλλά από το 92 δεν έχουμε τέτοιε τιμέ. Και το, είναι 15,6 ο περικοπή και όχι 38 όπως είπατε. Δεν υπάρχει όπως είπα από το 92 σύνδεση των πληρωμών του, ε, κοινού γεωργικού, της κοινής γεωργικής πολιτικής με τον πληθωρισμό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά εγώ σας το λέω. Τώρα, για την κατανομή των πληρωμών. Κοιτάξτε, υπάρχει ανώτατο όριο. Και όπως είπαμε υπάρχει ε, μείωση όσο αυξάνεται η, η, επιφάνεια που καλλιεργείται. Έτσι αποδεικνύουμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τις πληρωμές. Αλλά οι πληρωμές σήμερα βασίζονται στις επιφάνειες. Οι γεωργοί πληρώνονται με βάση τις ε, εκτάσεις και με βάση τους ορισμούς για το τι αποτελεί η γεωργική δραστηριότητα. Και έχουμε συγκεκριμένα μέτρα συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε τους ε, μικροκαλλιεργητές. Και ε, ελπίζω να υπάρξει στήριξη για να γίνει αυτό στη μεταρρύθμιση. Γιατί οι συνομοθέτε θα λάβουν την τελική απόφαση. Οι προτάσει Επιτροπή θα πρέπει να κρυθούν από εσά και ελπίζω να τι ε, στηρίξετε. Και ιδιαίτερα στι ανατολικέ χώρε που δεν δέχονται τον ορισμό αυτό ανωτά των τιμών για τι ενισχύσει και αναδιανομή αυτού που εξοικονομείται έτσι για την ανάπτυξη τη Δεν τα αναφέρατε όλα αυτά. Πρέπει να τα πω εγώ. 20% των δικαιούχων λαμβάνουν 84% των πληρωμών στη Ρουμανία. Ε, αυτό είναι το παλιό κομμουνιστικό σύστημα. Όπου υπάρχουν ε, όλοι αυτοί οι μεγαλογιοκτήμονε και οι μεγάλε εταιρείε που καλλιεργούν. Η πληρωμή ένα εκτάριο είναι πάνω από τον μέσο όρο. Από αυτά που λαμβάνουν αυτοί που έχουν 10 με 75 εκτάρια. Είναι θέμα. Είναι θέμα αλλά είναι ακούγεται σαν σύνθημα. Αν έχουμε ένα σύστημα, όπως όλοι πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε, όπου πληρώνουμε τους γεωργούς με βάση τις επιφάνειες που καλλιεργούν, εφόσον τις καλλιεργούν σωστά, να είναι πραγματικοί γεωργοί, τότε πρέπει να πληρώνονται σωστά. Ποιο θα την κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνουν οι γεωργοί. Για να επιτύχουμε και του άλλου στόχου. Σα προτείνω οι γεωργοί να το κάνουν αυτό. Τουλάχιστον εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Η Επιτροπή δεν έχει και τόσο πολλέ ε, εξουσίε για την ε, ε, χρήση γη. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αν το κράτη μέλη μα το δώσουν αυτήν την αρμοδιότητα, θα το κάνουμε. Αλλά δεν έχουμε αρμοδιότητε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε. Λοιπόν, για τη Σλοβακία. Ναι. Μα στείλατε, πρέπει να αναγνωρίσω, τον περασμένο Φεβρουάριο πολλή βιβλιογραφία για 13 περιπτώσεις όπου λέτε ότι υπάρχουν θέματα κακοδιαχείρισης, ε, εφαρμογή του κράτους δικαίου και απατών. Και μπερδεμένα όλα αυτά μαζί. Έκτοτε έγινε μία αστυνομική έρευνα και ασκήθηκαν διώξεις. Κάναμε ελέγχους από τότε που λάβαμε τα έγγραφα για να επαληθεύσουμε πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί πληρωμών και ελέγχου. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία ακόμη, αλλά σύντομα θα γίνει αυτό και θα σε ενημερώσουμε πλήρως για το τι πρόκειται να κάνουμε. Και το πρόγραμμα δράσης για τις άμεσες πληρωμές για την ε, Σλοβακία. Θα σε ενημερώνουμε για το πώς θα πάει. Η νέοι γεωργοί, βεβαίως, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί πρέπει να υπάρξει αλλαγή γενεών. Είναι ένα οριζόντιο θέμα όπως το προτείνουμε στη μεταρρύθμιση που δημοσιεύσαμε και στην πρόταση αυτή λέμε ότι δεν θα κρίνουμε κανένα στρατηγικό εθνικό πρόγραμμα εάν δεν περιέχει επαρκή μέτρα για την, ε, το πέρασμα της γεωργίας από τη μια γενιά στην άλλη. Και λέμε ότι μόνο 6% των δικαιούχων αυτή τη στιγμή είναι νέοι γεωργοί, δηλαδή κάτω των 40. Αυτό είναι ο ορισμός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν το δέχομαι. Αν θέλουμε να είναι πολύ πιο ζωηρή η γεωργική δραστηριότητα και η ζωή σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Το επιχειρήσαμε και προηγουμένως και οι συνομοθέτες δεν το δέχτηκαν. Και οι μεγαλύτερες οργανώσεις των γεωργών, που μπορεί στα διοικητικά τους συμβούλια να είναι πιο ηλικιωμένοι, πολλές φορές δεν θέλουν να στηρίξουν τους νεότερους. Αλλά θα πρέπει να το κάνουν περισσότερο από ό,τι κάνουν τώρα. Και μέσω της κοινή γεωργικής πολιτικής θα επιμείνουμε να γίνουν περισσότερα για τους νέους. Για την ΕΦΣΑ. Κοιτάξτε, δεν είμαι εμπειρονόμο για την ΕΦΣΑ. Δεν ξέρω τι προπολογισμό έχουν. Αλλά μπορούμε να σας στείλουμε απάντηση. Δεν είναι αρμοδιότητά μου. Αλλά επειδή έχω τόσο καλή διάθεση πάντα, θα παρακαλέσω τον συνάδελφο Ανδριουκάιτερ να σας στείλει απάντηση. Η βιολογική γεωργία. Ξέρετε, εγώ ήθελα να απαγορευτούν πλήρω τα φυτοφάρμακα για τα βιολογικά προϊόντα και οι πράσινοι με σταμάτησαν. Το ξέρετε αυτό. Επέμειναν. Επέμειναν. Επέμειναν δύο φυτοφάρμακα να επιτρέπονται για τη βιολογική γεωργία. Συγγνώμη σας το λέω. Αν είχε γίνει δεκτή η πρότασή μου, θα είχαμε ελάχιστα, βιολογικά, ελάχιστα φυτοφάρμακα συγγνώμη, στα βιολογικά. Αλλά οι πράσινοι αντιτέθηκαν, αλλά συγγνώμη, απέρριψαν την πρόταση της Κομισιόν να απογορευτούν πλήρως τα φυτοφάρμακα. Δεν με ικανοποιεί καθόλου η απάντησή σας. Εγώ είπα για τα, βιο, για τα φυτοφάρμακα, τα εισαγόμενα φυτοφάρμακα για όλα τα γεωργικά προϊόντα και γιατί γίνονται απάτες με τα εισαγόμενα βιολογικά γιατί δεν αναφέρεται ποιος τα παράγει και είναι αδύνατο να εντοπιστεί γιατί, γιατί κυρία Ριβασία, μα εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω με τα φυτοφάρμακα δεν έχω αρμοδιότητα από τι συζητήσει που έκανα για τη μεταρρύθμιση των βιολογικών. Ξέρω ότι οι πράσινοι ήταν κατά των προτάσεών μου. Πρόεδρο, αγαπητοί συνάδελφοι πραγματικά πρέπει να επικεντρωθούμε στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου. Δεν έχει αρμοδιότητα ούτε για τα τελωνιακά, ούτε για τους δασμούς, ούτε ε, για τα ερωτήματα που του απευθύνατε. Δεν είναι στον τομέα των αρμοδιοτήτων του αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να απευθυνθούμε στους αρμόδιους επιτρόπους για αυτά τα ερωτήματα. Είχαμε αποφασίσει στους συντονιστές το θέμα των ε, τελωνιακών ελέγχων να τεθεί στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας διότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις εισαγωγές όχι μόνο γεωργικών ε, προϊόντων αλλά και τα πλήγματα που δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τα οικονομικά της συμφέροντα μέσω των εισαγωγών. Απλά, ξαναλέω, δεν είναι ζήτηματα αρμοδιότητας του κύριου Χόγκαν θα τα ξαναδούμε αυτά τα ερωτήματα όταν θα συζητήσουμε ζητήματα τελωνιακών ελέγχων. Εκεί μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε και το θέμα των ε, μη επιτρεπόμενων φυτοφαρμάκων ε, στα κράτη-μέλη μας, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα ε, ενδιαφέρον ερώτημα. Όταν εντοπίζονται μη επιτρεπόμενα φυτοφάρμακα, τότε προφανώς και θα πρέπει να επισύρονται οι αναγκαίες εκείνες επιπτώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι και μέσω της ε, πολλαπλής ε, συμμόρφωσης η Γενική Διεύθυνση να μπορεί να λαμβάνει μέτρα σοβαρά όταν και όποτε πραγματικά διαπιστώνονται τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το εξετάσουμε ξεχωριστά, γιατί τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα πρέπει να δαπανώνται μόνο εφόσον υπάρχει τήρηση των οδηγιών και κανονισμών που έχουμε συναποφασίσει. Ο κύριος Χριστοφόρου ε, θα ήθελα να τοποθετηθεί. Ε, του δίνω λοιπόν τον ε, λόγο και ε, νομίζω ότι έχουμε τηρήσει και το χρονοδιάγραμμα. Κύριε Χριστοφόρου, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Ε, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για του λαού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γεωργικός τομέα και η αγροτική ανάπτυξη είναι από του πιο κρίσιμου τομεί είναι εκεί που κρίνεται και η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι χρειάζεται μεγάλη ικανότητα και δυνατότητα για να διαχειριστεί αυτόν τον τομέα της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης γιατί έχει να κάνει με χιλιάδες αγρότες, με χιλιάδες κόσμο που βρίσκεται στην Ήπεθρο με ιδιαίτερε συνθήκε, ιδιαίτερότητε, αλλά και αυξημένε ανάγκε από όλον αυτόν τον κόσμο. Είναι ακόμα δεδομένο ότι οι αγρότες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεινοπαθούν. Οι αγρότες που επιβίωσαν και πήραν ανάσα και βρίσκονται ακόμα όρθιοι και συνεχίζουν να σπούν αυτόν το ιδιαίτερα σκληρό επάγγελμα είναι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να διαλάθει τη προσοχή μας. Ανήκω και εγώ σε αυτούς που λυπάμαι που φεύγει ο αγαπητός Φιλ Χόκαν από την Ω Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτική ανάπτυξη. Γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπάρχει ένα αντικειμενικός κριτή σίγουρα θα πει ότι δεν λύθηκαν τα προβλήματα τη Γεωργίας και δεν μπορούν να λυθούν όλα. Είτε σε μια πενταετία είτε σε μια δεκαετία θα συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό τομέα. Πιστεύω όμω ότι ένα αντικειμενικός κριτή θα διαπιστώσει σε όλα τα επίπεδα ότι σε αυτήν την πενταετία ο επίτροπο και οι συνεργάτε του επιτέλεσα σημαντικών έργων και είχαμε βελτίωση σε όλα τα επίπεδα. Ένα βασικό πρόβλημα που είχε ο αγροτικό τομέα και η γεωργία μα ήταν η γραφειοκρατία. σω από του μοναδικού επιτρόπου που ήσυχοσε σημαία και έκανε πόλεμο ενάντια στη γραφειοκρατία για να εξυπηρετήσει του αγρότε μα, είναι ο επίτροπο σήμερα που βρίσκεται κοντά μα και οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και να τον συγχαρούμε για το σημαντικό έργο που υπήρξε και την βελτίωση. Δεν λύθηκε το πρόβλημα τη γραφειοκρατία. Όμω αυτό ο Επίτροπο έκανε το παν για να καθυποτάξει την γραφειοκρατία και να διευκολύνει του αγρότε. Για το μόνο που δεν ασχοληθήκαμε με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Με μία φράση του ελεκτικού συνέδριο είπε ότι όλε οι δράσει τη αγροτική ανάπτυξη έχουν υλοποιηθεί όπω έχουν σχεδιαστεί. Μακάρι σε όλου του επιτρόπου να υπήρχε αυτή η φράση μέσα στις, ως ρεζουμέ της εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου. Σημαίνει ότι τηρήθηκε με ακρίβεια αντικειμενικότητα και αξιοπιστία αυτών των οποίων εξαγγέρθηκε και πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί ο συγκεκριμένη επιτροπή έδωσε πραγματικά έναν αξιόπιστο δείγμα γραφής. Εμείς συμφωνούμε ακόμα και με τη φιλοσοφία του Επιτρόπου και πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έπρεπε να συμφωνούν ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε τον κόσμο αυτό κι αν είναι κάτι φιλολαϊκό που έπρεπε από όλε τι ομάδε να χαιρετιστεί. Ότι αυτή η φιλοσοφία ότι χρειάζεται ένα νέο σύστημα προληπτικού ελέγχου και ότι ο στόχο μα δεν είναι να κυνηγάμε τον αγρότη, να κυνηγάμε τον γεωργό. Εκεί και όπου υπάρχει απάτη να είμαστε σκληροί και αμήλικτοι, αλλά η πρόθεση δεν είναι να ποινικοποιούμε του αγρότε και του γεωργού και να του τρέχουμε πίσω για να ανακαλύψουμε αν είχαν έναν human error, όπω λέγεται προηγουμένω. Και τελειώνοντα, θέλω να πω ότι θα ήταν σημαντικό να μα πει ο κύριο Επίτροπο πώ διατέθηκαν στου αγρότε μα όλα αυτά τα κονδύλια. Και κυρία Πρόεδρε, επιστρέψτε με, επειδή κάνατε αναφορά στην Κύπρο, να πω ότι υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να γνωρίζει η Επιτροπή μα, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι. Ότι σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν οι μοναδικοί χιλιάδε γεωργοί που δεν παίρνουν καμιά νεκταρική επιδότηση. Είναι οι πρόσφυγε γεωργοί τη Κύπρου, οι οποίοι διαθέτουν χιλιάδε εκτάρια γης που δεν μπορούν να τα καλλιεργήσουν γιατί τους εμποδίζει ο στρατός κατοχής. Και είναι τεράστια δικία το ότι θεωρείται όλη η επικράτεια ευρωπαϊκού έδαφος, δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν πήραν ούτε ένα σεν ενώ είναι αγρότες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχω και εγώ ένα τελείως διαφορετικό ερώτημα να θέσω στον ε, Επίτροπο αν και γνωρίζουμε ότι δεν είστε αρμόδιος για τα φυτοφάρμακα. Ξέρουμε όμως ότι όταν χρησιμοποιούνται παράνομα φυτοφάρμακα ε, μπορούν να διατεθούν με μικρότερο κόστος προϊόντα στην αγορά, κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε στρέβλωση της αγοράς. Η δική σας Γενική Διεύθυνση έχει λάβει γνώση τέτοιων πρακτικών, ιδίως σε χώρες όπου η διοίκηση έχει προβλήματα. Εκεί όπου οι έλεγχοι δεν γίνονται με τον προβλεπόμενο τρόπο, δεν γίνονται με τον ενδειγμένο τρόπο. Υπάρχουν ε, πληροφορίες ότι υπάρχουν τέτοιες ε, παρατυπίες. Υπάρχουν ε, πληροφορίες, υπάρχουν έρευνες ενδεχομένως που βρίσκονται σε εξέλιξη σε κρατημέλη όποτε εμφανίστηκαν τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί είναι και πάντοτε μια αλυσίδωτη αντίδραση. Μπορεί κάποια άλλη ε, ε, υπηρεσία να το ξεκινάει, την έρευνα, όμως τελικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και για τις ε, ε, επιχορηγήσεις με βάση την έκταση. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα. Πείτε μας. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ τον κύριο Χριστοφόρο για τα καλά του λόγια. Νομίζω ότι έχει τίποτα άλλο να με ρωτήσει. Τέλος πάντων, ευχαριστώ για όσα είπε. Πρόεδρε, το θέμα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά χρειάζεται περισσότερη συνεργασία περισσότερων γενικών διευθύνσεων. Η Γεωργία, ποιότητα των τροφίμων, εισαγωγές, εναρμόνιση, προτυποποίηση. Αυτά είναι στο νέο μου χαρτοφυλάγιο Άρα είναι και θέμα εμπορίου. Εκτό από γεωργίε. Οπότε θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό και πάντοτε και των πολιτών και οι φορείς μας ενδιαφέρουν το πώς θα γίνει καλύτερη συνεργασία, να υπάρχουν κοινά πρωτόκολλα και τα κράτη-μέλη να έχουν κατευθυντήριες για ελέγχους. Υπάρχουν, αλλά συμφωνώ. Γιατί δεν είναι οι σχετικοί κανόνες εναρμονισμένοι. Οπότε θα το κοιτάξω και θα σας πω. Γι' αυτό που είπατε, γι' αυτό που ρωτήσατε, εύκολη απάντηση δεν υπάρχει τώρα. Δεν έχουμε τον αρκετό συντονισμό. Α, με την ε, νέα Κυπρία Επίτροπο που θα έχει το σχετικό χαρτοφυλάκιο και ε, την Πολωνία τον Πολωνό ε, θα το κοιτάξουν και θα σας πούμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το γεγονός ότι απαντήσατε διεξοδικά τις ερωτήσεις μας. Εγώ ως εισηγήτρια βεβαίως θα επιτρέψω τον εαυτό μου να, ξανα, να επανέλθω ε, στα ερωτήματά μου. Θέλω να μιλήσω και για τα όσα είπε ο κύριος Χριστοφόρου. Το πρόβλημα της Βορείας Κύπρου δυστυχώς δεν είναι γεωργικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα διεθνούς δικαίου ε, μεταξύ δύο κρατών όπου ένα ε, τμήμα του ενός κράτους βρίσκεται υποκατοχή. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε την πλήρη υποστήριξή μας κύριε Χριστοφόρου διότι ο προϋπολογισμός προβλέπει και δαπάνες και για αυτόν τον ε, σκοπό και καταβάλουμε προσπάθειες τουλάχιστον ε, στο μέλλον ε, τα ζητήματα αυτά να τα χειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο. Βεβαίως δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός να υπερβεί αυτή η διχασμένη χώρα τα προβλήματά της. Και ως Γερμανίδα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ξέρω πραγματικά πόσο επώδυνη είναι η κατάσταση αυτή. Κύριε Επίτροπε, ε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν σας αποχαιρετώ οριστικό. Θα σας ξαναδούμε ως Επίτροπο για ζητήματα εμπορίου. Και εκεί βεβαίως θα σας βομβαρδίσουμε πια με άλλα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ πάντως για το γεγονός ότι ήσασταν εδώ και για, την, για τις εξαιρετικές απαντήσεις που μας ε, δώσατε. Ευχαριστώ. Θέλω απλώς να πω στον κύριο Χριστοφόρου ότι ε, ως Επιτροπή είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 20% των γεωργών στην Κύπρο λαμβάνουν το 75% των επιχορηγήσεων. Αυτό δεν συμβαίνει ε, συχνά σε μια χώρα με, με πολλούς μικρούς ε, γεωργούς. Το ίδιο συμβαίνει και στην ε, Ρουμανία. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στη διάρκεια αυτής της θητείας μου. Ξαναλέω, ότι έγιναν πολλά, σημειώθηκε πρόοδο, αλλά είναι αυτή η κλασική περίπτωση που λες ότι πολλά έγιναν, αλλά που θα μπορούσαν να είχαν γίνει και πολλά ακόμα και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα Θέλω να ευχαριστήσω το επιτελείο μου, τους ανθρώπους της Γενικής Διεύθυνση Γεωργία, τον Γενικό Διευθυντή που έκαναν ό,τι καλύτερο προκειμένου να εφαρμόσουν τα όσα έχουν συναποφασίσει οι συνομοθέτες με ταυτόχρονο σεβασμό στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Να ευχαριστήσω επίσης και το ελεγκτικό συνέδριο που τα τελευταία χρόνια είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Δεν ξέρω τι έγινε, πάντως δεν, δεν ξέρω τι έγινε με το χέρι σας κύριε Μιλιώνη. Εγώ δεν το έκανα σε κάθε περίπτωση. Ε, ο Επίτροπος ε, διαψεύδει τη φήμη ότι πριν τη συνεδρίαση έσπασε το χέρι του κυρίου Μιλιώνη. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν ε, την Επιτροπή σας για όλη τη στήριξη που μου παρήχατε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Επίτροπε, να είστε βέβαιος ότι θα επανέλθουμε το ζήτημα ε, των ενισχύσεων σε μεγάλους μικρούς γε, γεωργούς και τη μετακίνηση που υπάρχει από τους μικρούς στους μεγαλύτερους γεωργούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Μιλιώνη, το μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Προσβλέπουμε στην μελλοντική συνεργασία και μαζί σας και βεβαίως και με τον ε, μελλοντικό επίτροπο και με τον παλιό επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν, αλλά σε νέες ευθύνες, σε νέους τομείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

May uh, Πρόεδρος, παρακαλώ. Παρακαλώ, συνάδελφοι. Και οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Συνεδρίου να αποχωρήσετε ησύχως. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο και το Επιτελείο του, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γιατί έχουμε άλλα δύο θέματα. Έχουν να κάνουν με κάποια ζητήματα επί των οποίων τα μέλη, οι εκπρόσωποι τέλο πάντων του συνεδρίου θα μας τα εξηγήσουν. Υπάρχουν τέσσερα θέματα όσον αφορά την επίκριση των επιδόσεων για την συνοχή και θερμά καλωσορίσματα στην πρώην συνάδελφο και νυν έμπειρη ε, σύμβουλο πολιτικού Συνεδρίου. Η κυρία Πανόβα. Uh, forward to listening to you uh, and uh, to... Και να μας πεις, συνάδελφε, αυτά τα οποία αφορούν την ε, επίτευξη επιδόσεων στην συνοχή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι ε, βουλευτέ. Είναι μεγάλη μου χαρά που τώρα επανέρχομαι στην Επιτροπή Ελέγχων των Προπολών για πρώτη φορά μετά την συγκρότηση του νέου κοινοβουλίου. Και ήρθα σήμερα να σας παρουσιάσω αυτό το ενημερωτικό έγγραφο όσον αφορά τις επιδόσεις στην συνολική και το πρώτο που έχω να σας πω ότι δεν πρόκειται για έκθεση οικονομικού ελέγχου είναι απλώς ενημερωτικό. Ποια είναι η διαφορά? Ότι Αυτά τα ενημερωτικά δεν περιέχουν αξιολογήσεις κατόπιν ελέγχων και συστάσεις. Ο στόχος είναι η κωδικοποίηση πληροφοριών που ήδη υπάρχουν και έτσι να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε την ε, προβληματική για τα επίκαιρα. Έχουμε ένα σωρό εκθέσεις 69 συνολικά, αυτές που έχουν γίνει όσον αφορά τη συνοχή την τελευταία δεκαετία. Αυτές οι πληροφορίες εδόθησαν και επαληθεύτηκαν και από μελέτες των θεσμικών οργάνων αλλά και εξωτερικών όπως ο, ο ΣΑ. Στόχος ήταν να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής επικεντρώνεται στις επιδόσεις και όχι στην συμμόρφωση. Αυτό ήταν η αποδόση σε όλες τις ε, εκθέσεις. Θέλουμε εκεί να έχουμε πιο σφαιρική ενημέρωση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ε, περίοδο του, ε, του πλαισίου ε, σε σχέση με την ε, επόμενη. Και έχουμε τέσσερι ε, κατευθυντήριε, δέκατε συγγνώμη κατευθυντήριε αρχέ που χρειάζονται για να μπορέσουμε να είναι πιο αποδοτική η πολιτική συνοχή. Είναι τα βασικά θέματα τα οποία επισημάνομαι και έτσι μπορούμε να αξιολογήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, κοιτάξτε τώρα εδώ, σε, αυτό, σε αυτή τη διαφάνεια, τι γίνεται με τον όλο κύκλο και αυτές τις καθημερινές ε, αρχές. Έχουμε πέντε ε, φάσεις σε αυτή τη διαχείριση και όλα τα και όλες τις ε, αρχές και υπάρχει και βέβαια η βιωσιμότητα που είναι η αρχή που ε, τις διαπνέει όλες τις άλλες, μην πούμε τις 14 αρχές μία-μία, ας τις ε, ομαδοποιήσουμε ε, επί τη βάση αυτού του κύκλου υλοποίησης. Οπότε η πρώτη φάση είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, εδώ έχουμε δύο σχετικές άρχες, πρώτα-πρώτα το ότι χρειάζεται να υπάρχει κάποιο στρατηγικό όραμα, στρατηγική οπτική, και αυτά τα βλέπετε στην αρχή αυτής της ε, ενημέρωσης. Εδώ με αυτά τα χρώματα. Εδώ το φανάρι ας το πούμε. Το φανάρι είναι κόκκινο. Και βλέπουμε τι γίνεται στην επόμενη περίοδο. Είναι για από αυτό κάτι σημαίνει. Και η εκτίμησή μας είναι ότι η κατάσταση είναι κάπως χειρότερη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τώρα έχουμε πάει στο κίτρινο και ο βασικός λόγος είναι οι στρατηγικές του 2020 τώρα ολοκληρώνονται, αλλά ακόμη δεν έχουν υποκατασταθεί από άλλες. Οπότε βλέπουμε ότι δεν έχουμε κάποιο όραμα στρατηγικό σε σχέση με το όραμα 2020 ε, και τη στρατηγική της Λισαβόνας και έτσι δεν έχουμε κάποιο σχήμα του τι θέλουμε να πετύχουμε. Άλλη γενική αρχή είναι το πώς γίνεται η χορήγηση των πόρων στα κρατή-μέλη. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ενημερωτικό πιο εντελεχές που λέει ακριβώς τι γίνεται με τη διαδικασία της χορήγησης των πόρων. Και εδώ το φανάρι είναι κίτρινο. Πάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια ε, και φάση του κύκλου είναι ο προγραμματισμός. Εδώ ετοιμάζουν τα κράτη-μέλη το πώς ε, προτίθενται να αναλώσουν τα κονδύλια. Εδώ έχουμε τέσσερις καθυντήριες και μπορεί να δείτε από την αξιολόγησή μας ότι εδώ είμαστε πιο θετικοί σε σχέση με πριν. Ε, δύο φορές έχουμε το πράσινο εδώ σε δύο σημεία και σε σχέση με την τελευταία κατευθυντήρια ακόμα υπάρχει περιθώριο για περισσότερα κίνητρα στην επίδοση για το τι γίνεται με την χρηματοδότηση. Έχει κάποιους μηχανισμούς η Κομισιόν στο τέλος αυτής της περίοδου. Περιορισμένα τα αποτελέσματα και έχουμε τώρα τις προτάσεις για την επόμενη περίοδο. Οπότε Ούτε εδώ όσον αφορά τους στόχους επιτύχους αποτελεσμάτων δεν έχουμε τα ε, επιθυμητά από τις ε, χορηγίες. Στην επόμενη φάση έχουμε τη φάση της υλοποίησης από τα κράτη-μέλη. Όπως είπαμε εδώ έχουμε τρεις βασικές κατευθυντήριες αρχές και εδώ η γενική κατάσταση είναι λιγότερο ρόδινη. Ο πάντως είναι ε, καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν και για την επόμενη περίοδο έχουμε την καθημερινή 9 αναθεώρηση των προγραμμάτων πριν είχαμε δύο κίτρινα, τώρα έχουμε επιδείνωση και τα προγράμματα των κρατών μελών ίσως αναθεωρηθούν, αλλά δεν έχει μελετηθεί η επίπτωση στην επίδοση. Το νομοθετικό πλαίσιο τώρα το 2020 θα πρέπει να δούμε αν ε, δικαιολογούνται οι αλλαγές στα προγράμματα για επιτευξή των στόχων μαζί με, τα, με τους κανόνες σε σχέση με τους δείκτες. Για την περίοδο 2027, ε, εδώ πέρα υπάρχουμε, ε, έχει υποχρεωτική ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν είναι σαφές το πώς θα αξιολογηθεί η επίδοση και τα κράτη-μέλη πώς θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την χορήγηση αφού δεν θα έχουμε ε, θεώρηση των αποτελεσμάτων. Τώρα έχουμε έλεγχο, εποπτεία και τις σχετικές εκθέσεις, αναφορές και εδώ είμαστε στο κίτρινο. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τις τρεις ε, εν προκειμένου εξεταζόμενε περιόδου. Ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι η έκθεση και η υποβολή των εκθέσεων εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων. Τα περισσότερα έρχονται από τα κράτη-μέλη πριν διαβαστούν στην Κομισιόν και εδώ υπάρχουν μειονεκτήματα ποιοτικά. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Τα λέμε στις εκθέσεις μας, δίνουμε και κάποια παραδείγματα στο ενημερωτικό αλλά και το θέμα της ανεργίας των νέων ή της απασχόλησης των νέων, παιδεία, κατάρτιση, εκπαίδευση τέλο πάντων κατάρτιση. Σε επόμενη περίοδο εδώ θα είπαμε ότι η Επιτροπή θα το αντιμετωπίσει, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την ποιότητα των ε, δεδομένων. Τελευταίο, αλλά σημαντικό πολύ βασική φάση αυτού του κύκλου είναι η αξιολόγηση. Εδώ έχουμε μία κατευθυντηριά αρχή, αλλά εδώ λέμε ότι είναι οριζόντια σημασία της ε, βιωσιμότητας, κίτρινο εδώ, και για τις τρεις αξιολογηθήσεις περίοδους. Στο σύνολό τη η Επιτροπή έχει ένα καλοσχεδιασμένο σύστημα αξιολόγησης και αναθεώρησης σε σχέση με τα κρατή μέλη, τα περισσότερα, και το 18 το σύστημά μας όσα είπε ότι είναι τέταρτο ε, εν μέσω των υπολείπων μελών του όσα είπαμε για τη χρησιμότητα της αξιολόγησης ε, εδώ κίτρινο δεν χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις για την λήψη αποφάσεων πολλές φορές ε, δεν έρχονται έγκαιρα ή δεν ε, αρκούν οι χρησιμοποιούμενες αποδείξεις, τα στοιχεία τέλο πάντων. Τώρα, ε, βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες ειδικέ εκθέσεις που επισημαίνουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν για τη βιωσιμότητα σε διάφορες φάσεις, στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης. Και εδώ σας ε, δίνουμε μία εικόνα ε, της γενικής αξιολόγησης και για τις 14 διευθυντήριε ε, αρχές και για τις τρεις περιόδους πολιετών πλαισίων. Βλέπετε τι γίνεται μεταξύ πρώτης και τρίτης ε, περίοδου που έχουμε πολλά κόκκινα, κυρίω 7 ε, με 13 και περισσότερες βελτιώσεις συνέβησαν κατά την τρέχουσα περίοδο 14 με 20 μικρή ή καθόλου βελτίωση ε, σε σχέση με δεύτερη και τρίτη περίοδο. Πώς βλέπετε και αυτό, ε, ακριβώς όπως τα είπαμε πέρσι για τις προτάσεις της Κομισιόν, όπου εκεί λεπτομερώς είχαμε εξεταστεί νομοθεσία, δεν ε, ασχολούμασταν με τις επιδόσεις. Αυτά ήθελα να σας πω δύο λίγο. Πρόεδρε, ευχαρίστως να απαντήσω σε ερωτήσεις και να ακούσω παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε εδώ το Διευθυντή της Κομισιόν. Αν θέλει το λόγο. Και κατόπιν ο κύριος Σανιέτσι απευθείας, ο συγκητή μας. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Ιβάνοβα και το συνέδριο για αυτό το έγγραφο. Χαιρόμαστε που το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει ότι το νομικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχει εξελιχθεί θετικά, είναι πιο εστιάζει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχής έχει το πιο πλήρες ε, πλαίσιο πολιτικής από όλες τις ενωσιακές πολιτικές. Για παράδειγμα, κάναμε αυτή την ε, αξιολόγηση πρόσφατα απόδοσης όπου εξετάμε, ε, εξετάζουμε αν επέτυχαν τους στόχους τα προγράμματα. Είχαμε έξι, προγρά... έξι στόχους στην αρχή της ε, περίοδου προγραμματισμού και τα προγράμματα που το έχουν επιτύχει θα πάρουν ένα 6% μπόνους και τα προγράμματα που δεν ε, έχουν επιτύχει τους στόχους θα έχουν 6% πρόστιμο. Άρα 3 δις θα πάνε από τα καλύτερα, μάλλον αντίστροφα, από τα χειρότερα στα καλύτερα προγράμματα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μας ενδιαφέρει. Να επιτυχάνουμε αποτελέσματα αυτά για τους συμπολίτες μας. Να δώσω και εδώ μερικά στοιχεία. Το πρώτο είναι Μόλις ε, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη περίοδος προγραμματισμού και τι είδαμε. Δημιουργήσαμε μέσω ενωσιακής χρηματοδότησης πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και ενισχύσαμε την ε, παραγωγικότητα πάνω από 400, σε πάνω από 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα προφανώ. Αυτό είναι πάντα ο στόχο μας. Και εδώ υπάρχουν κάποια σημεία όπου διαφωνούμε με τα πορίσματα του συνεδρίου. Αντίθετα με αυτά που προτείνει το συνέδριο. Νομίζουμε ότι το μελλοντικό μας νομικό πλαίσιο είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ συνέχειας και απλούστευσης. Δηλαδή, τα καλά τα κρατάμε, τα άλλα τα πλουστεύουμε. Να αναφερθώ σε θέματα που έθιξε και το συνέδριο. Το μελλοντικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής θα εστιάσει σε πέντε πυλώνες. Πιο ευφυή Ευρώπη, πιο πράσινη Ευρώπη, πιο κοινωνική Ευρώπη, πιο συνδεδεμένη Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Αυτοί οι πέντε στόχοι νομίζω ότι εντάσσονται πλήρω στην ευρύτερη ενωσιακή πολιτική. Όλα αυτά θα τα συνδέσουμε πιο πολύ, την πολιτική συνοχή δηλαδή, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα έχουμε λοιπόν μια πιο πλήρη γνώση των προβλημάτων που έχουμε για τις δημόσιες επενδύσεις, τις δημόσιες δαπάνες για παράδειγμα και αυτό θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν από τα προγράμματα, τα μελλοντικά προγράμματα συνοχής που θα τα επιτηρεί συνεχώς η Επιτροπή. Επίσης, αυτό που θα διατηρήσουμε και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, γιατί το διαπιστώσαμε στην τρέχουσα, είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δημιουργήσουν το καλύτερο πλαίσιο για να έχουν αντίκτυπο ή επενδύσεις. Και στο μέλλον, λοιπόν, θα πρέπει να είναι κάποιες διευκολυντικές ε, συνθήκες για τις δημόσιες προμήθειες, τις κρατικές βοήθειες, αλλά και για παράδειγμα οι επενδύσεις για το κλίμα, οι επενδύσεις συνοχής θα πρέπει να βοηθούν τη γενικότερη πολιτική των κρατών μελών για το κλίμα στα πλαίσια της επίτευξης των στόχων του 2030. Επίσης, Νομίζω ότι είμαστε πιο στοχευμένοι στην επίτευξη αποτελεσμάτων, στην υψηλή απόδοση. Πάνω από 6% της χρηματοδότησής μας δόθηκε, ήδη όπως σας είπα, και στο μέλλον θα κάνουμε Το 2026 και το 2027 για τις ε, ε, πληρωμές εκείνης της εποχής θα χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες το 2024 και θα θέσουμε το ερώτημα εάν πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό η χρηματοδότησή μας με βάση την απόδοση των προγραμμάτων. Και κάτι άλλο που λέει και το συνέδριο. Η σημασία το επόμενο νομικό πλαίσιο να εγκριθεί τάχιστα. Διότι αλλιώς θα έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Και αυτό θα επιδράσει και επί των επενδύσεων, άρα θα επηρεάσει και την ευημερία των συμπολιτών μας. Οπότε κάνω έκκληση. Κάντε ό,τι μπορείτε παρακαλώ για να εγκριθεί τάχιστα το νομικό πλαίσιο. Σε συνεργασία πάντα βέβαια με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λίγο στον κύριο Τσαρνέτσκι, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ιβάνοβα, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κυρία Ιβάνοβα, για το εξαιρετικό αυτό ενημερωτικό σημείωμα που περιέχει πολύ σημαντικές πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κάποια αριθμητικά στοιχεία για την πολιτική συνεχή. Σε διάφορες περιπτώσεις, στη διάρκεια της τελευταίας ε, θητείας της Κομισιόν, με τον ε, Επίτροπο Αρμόδιο για τον Προπολογισμό, τον κύριο Έτιγκερ, ε, υπόθηκε ότι η σημασία των επιστροφών των δαπανών του προϋπολογισμού θα πρέπει να κατευθεί κατά κύριο λόγο στους καθαρά συνεισφέροντες. Η Γερμανία ωφελείται από χρήματα που δαπανώνται σε χώρες συνοχής μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της. υλικά, κατασκευαστικός τομέας, ε, βαρύς ε, εξοπλισμός και στην τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ECR, η δική μου πολιτική ομάδα, απίφθινε και γραπτό ερώτημα προς την Κομισιόν με το αίτημα να γίνουν μελέτες όσον αφορά το θέμα αυτό. Η Επιτροπή διεξήγαγε μια τέτοια μελέτη και σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, σύμφωνα με τη ε, μελέτη του, του Πολωνικού Υπουργείου, κάθε ευρώ που δαπανι, δαπανάται ε, στην Πολωνία στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η Γερμανία ωφελείται ε, κατά 0,72 του ευρώ ε, μέσω προϊόντων που ε, παρέχει ε, στην Πολωνία. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση με βάση αυτά τα στοιχεία. Μπαίνοντα σε πιο λεπτομερή θέματα, θέλω να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα. Οι στόχοι στρατηγική θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Σύμφωνα με το συνέδριο, οι στόχοι στρατηγική δεν ήταν πάντοτε ε, οι ενδεδειγμένοι ή δεν λάμβαναν υπόψη την ε, διαθέσιμη χρηματοδότηση. Επίση, οι δράσει θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με το συνέδριο, οι δράσει αυτέ πολύ συχνά δεν συνδέονταν ξεκάθαρα με τους στόχους που εξυπηρετούσαν ή δεν επικεντρώνονταν επαρκώς στα αποτελέσματα. Επίσης, οι πληροφορίες επιδόσεων που κοινοποιούν τα κράτη-μέλη ε, προς την Κομισιόν θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και θα πρέπει να δημιουργούνται μόνο όταν χρειάζεται. Για παράδειγμα, για τη λήψη των μέτρων ή την υποστήριξη τη εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά που αναφέρονται στο έγγραφο και πολύ, με πολύ μεγάλη χαρά ε, θα περιμένω να παρακολουθήσω την ε, συζήτηση. Α, και να κάνω και μια ακόμη παρατήρηση. Συμπληρωματική. Με χαρά διάβασα ότι το 2018 η ε, ΩΣΑ κατέταξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέταρτη χώρα ε, στη διενέργεια εκτονιστέρων εκ ελέγχων. Αυτό θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε βεβαίως και την προέλευση των ε, προϊόντων ε, με θετικό τρόπο. Κυρία Πένκοβα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την λεπτομερή παρουσίαση. Το ενημερωτικό αυτό σημείωμα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο όσον αφορά τις κατευθύνες γραμμές που αναδεικνύονται μέσα σε αυτό και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι διαπιστώνεται μια γενική πρόοδος, ε, μια μετατόπιση προς τις επιδόσεις. Βεβαίως διαπιστώνουμε όλοι ότι χρειάζονται ακόμα περαιτέρω ε, βελτιώσεις και το συνέδριο σωστά ε, τονίζει την ανάγκη ενίσχυση τη αποτελεσματικότητα και τη αποδοτικότητα ε, τη πολιτική συνοχή. Σα ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το σημείο. Θέλω να απευθύνω και κάποια ερωτήματα στο ελεγκτικό συνέδριο και στου εκπροσώπους τη Κομισιόν. Πρώτο ερώτημα. Δεδομένου ότι τονίζουμε τη σημασία τη σύνδεση των επιδόσεων με τι δαπάνε του προπολογισμού. Το υποχρεωτικό αποθεματικό επιδόσεων που υπήρχε στην προηγούμενη περίοδο ε, πλέον αφαιρείται για την επόμενη προγραμματική περίοδο από την Κομισιόν. Και ανταυτού η Κομισιόν επιδιώκει να κάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση Το 2025 συγκεκριμένα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποιον ακριβώς τρόπο η αναθεώρηση αυτή θα διεξαχθεί και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι θα μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεύτερο ερώτημα και τελευταίο από πλευράς μου. Οι αιτήσει εκθέσει μετά το 2018 έχουν αλλάξει και πρέπει πλέον να δηλώνεται ότι η... τα στοιχεία ε, είναι σωστά και όσον αφορά τις επιδόσεις και όχι μόνο όσον, αφορά εκείνα που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Πώς αυτή η υποχρέωση θα εφαρμοστεί στην πράξη στο μέλλον. Δεδομένου ότι και το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει, έχει, έχει δηλώσει ότι δεν έχει ακόμα εξετάσει σε βάθος ε, αυτήν την ε, ένταξη των ε, στοιχείων και των δεδομένων επιδόσεων. Θα μπορείτε εσείς να τα εντάσετε όλα αυτά στο, στην ετήσια έκθεση που συντάσσετε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ivanova, and also the representative of the... Ευχαριστούμε και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, διότι μας είπε για την ενδιαφέρουσα έκθεση μας έκανε κάποιες παρατηρήσεις για όλους μας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος της είναι η εξάλληψη των ανισοτήτων στις περιφέρειες, εξισορρόπηση της ανάπτυξης οικονομικής πλευράς και άλλες και βέβαια χρειάζεται να έχουμε θετικές αλλαγές επί τη βάση του κριτηρίου της επίτευξης επιδόσεων γιατί προς το παρόν δεν πετυχαίνουμε με τους πόρους της συνοχής αυτό που θέλουν πολλές φορές κάνουμε το αντίθετο του σκοπημένου. Στην Ουγγαρία πολλές φορές αυξάνονται οι ανισότητες γιατί πάρα πολλοί ε, μειονεκτούντες δεν έχουν πρόσβαση στη, στα κονδύλια τα κοινωτικά επίσης δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα για τις δέουσες επιδόσεις οπότε σας ερωτώ με τι μέσα και εργαλεία θα δώσετε κίνητρα στα κρατημέλη για καλύτερες επιδόσεις και κυρίως να τους δώσετε κίνητρα για να υπάρχει με ίσο τρόπο κάλυψη όλων των γενικών ομάδων και ιδίως των μειονεκτούντων. Επίσης η εμπειρία μας λέει ότι η χρήση των κονδυλίων πολλές φορές γίνεται με πολιτικά κριτήρια. Η Ρέγγιο πρόσφατα κατέληξε στο ότι στην Ουγγαρία με υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων πολλές φορές οι αποφάσεις ήταν πολιτικοποιημένες, δεν υπήρχαν σαφή κριτήρια επιλογής ούτε υπήρχε κάποιο είδους πρόβλεψη για 11 μέσα πρόσφυγης. Οπότε, έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλει να πετύχει με τους πόρους της συνοχής. Πολλές φορές, οι στρατηγικοί στόχοι δεν μεταφράζονται σε επιχειρησιακούς, λειτουργικούς στόχους. Πολλές φορές οι στόχοι παραμένουν σε επίπεδο πολιτικών φιλοδοξιών. Λέμε ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν μπορούμε να δούμε τι ανάγκες έχουν εντοπιστεί στα κράτη-μέλη, άρα οι κανόνες και οι στόχοι είναι ασαφείς, αλλά και οι κανόνες, οι πραγματικές ανάγκες των κρατών δεν έχουν την υπόψη. Εσείς πώς πιστεύετε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των στόχων και μεταξύ τρόπων να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες κατά των μελών και να μην έχουμε κίνδυνο παρέμβαση της κυβέρνησης που να ασκεί την πολιτική μόνο με βάση πολιτικά κριτήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να δώσω και πάλι το λόγο στην ε, κυρία Ιλιάνα Ιβάνοβα για να τοποθετηθεί σε αυτά που είπε ε, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ε, βουλευτές για τις αξιόλογες ερωτήσεις για να δούμε αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος εισηγητής τον οποίο και ευχαριστώ κύριε Τσαρνέσκη πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά του στρατηγικού στόχου που θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί συμφωνώ 100% μέσα γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα οριζόντιο, εγκάρσιο αφορά πάσα έκθεση μας να και εγώ ήμουν εισηγήτρια για την απασχόληση των νέων και ο στόχος ήταν να πετύχουμε κάθε νέος να έχει εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία, δουλειά. μόλι μπει στην ε, αγορά απασχόληση. Δεν ήταν ρεαλιστικό αυτό σε υπόσχεση και η Κομισιόν το είχε αναγνωρίσει στην Λευκή Βίβλο. Υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ προσδοκιών και δυνατοτήτων Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Άλλο παράδειγμα για την ευρυζωνικότητα, τα νοικοκυριά. Τους υποσχεθήκαμε να έχουν ευρυζωνικότητα γρήγορη κάποια στιγμή. Ε, αυτά δεν είναι ρεαλιστικά. Από την αρχή είναι προφανές ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα, παρόλα αυτά όμως τα υποσχόμαστε. Ε, αυτό είναι το μήνυμα. Να είμαστε ρεαλιστές από την αρχή. Τι μπορεί να πετύχεις, και τι μπορείς να υποσχεθείς. Και έτσι στο μέλλον να το αποφύγουμε αυτό. Ιδίω όσον να είναι εγγύηση για την προσχολή των νέων και όλα αυτά για τους νέους. Οπότε αυτό φέρνει μια, μια απογοήτευση και μετά άντε να ξαναβρεις την εμπιστοσύνη τους. Τα είπαμε και αυτά και στον ημερωτικό. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα από όλες τις ειδικέ μας ε, εκθέσεις τόσα χρόνια. Για το αποθεματικό επιδόσεων. Συμφωνώ με αυτό που είπατε, το είπαμε και στη γνωμοδότηση όσον αφορά τον κανονισμό και των διατάξεων. Θεωρούσαμε ότι δεν είναι καλή ιδέα να καταργηθεί αυτό το μέτρο. Όμω θα εξηγήσει καλύτερα μα η όσον αφορά τι αιτήσει δραστηριότητε και τι εκθέσει. Σας είπα, αυτό που τώρα εξετάζουμε είναι κάτι που ανακεφαλαιώνει την προηγούμενη δουλειά ενημερωτικά. Και όταν το συντάξαμε, δεν μπορέσαμε να καλύψουμε αυτό το θέμα, αλλά στην επόμενη της έκθεση θα το καλύψουμε. Και σας ενημερώνω ότι του χρόνου σχεδιάζουμε μια ειδική έκθεση ακριβώς για κίνητρα και επιδόσεις. Αυτό φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει και του χρόνου θα αρχίσουμε την σύνταξη αυτού του εγγράφου. Τώρα, για το πώς θα βρεθεί η δέουσα ισορροπία, δύσκολο. Τα ακούω όλα μου τα χρόνια. Και εδώ στην Επιτροπή και αλλού. Και είναι σημαντικό να απασχίσουμε, να βρούμε αυτή την ε, ισορροπία. Γιατί καλή η απλούστευση, αλλά έχει κόστος, έχει τίμημα και το θέμα θα γίνει με την, επίδοση επιδόσεις. Τώρα για τον κανονισμό των κοινών διατάξεων τα λέει το ενημερωτικό ότι οι επιδόσεις είναι μια σοβαρή πτυχή Όπως έχει εξελιχθεί η πολιτική συνοχή, έχει βελτιωθεί, αλλά θα πρέπει ο κόσμος να νιώσει τα αποτελέσματα. Πώς, πού θα βρούμε τη σωστή ισορροπία λοιπόν. Προσπάθεια που συνεχίζεται. Ελπίζουμε να λυθούν υπόψη οι συστάσεις μας από την Κομισιόν. και βλέπουμε τις βελτιώσεις, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ θερμά. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ το μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα. Και να τα ξαναπούμε σύντομα. Και τώρα, το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη Ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την απαλλαγή 2018 για την μετώπιση των απατών στην συνοχή. Πρέπει να ενισχύσουμε τον εντοπισμό, την ανταπόκριση και τον συντονισμό. Αυτό αναφέρθηκε συγκεκριμένα όταν εδώ ο Πρόεδρος λένε είπε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την τεχνική βοήθεια και για την επιχειρησιακή πλευρά. Λοιπόν, ο κύριος Γκρέτεν. Έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά Χριστοφόρου. Κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που μπορώ να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση για την αντιμετώπιση της απάτης στις δαπάνες συνοχής. Μερικά στατιστικά στοιχεία. Μεταξύ του 2013 και 2017 η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη εντόπισαν πάνω από 4.000 ενδεχόμενα κακόβουλες παρατυπίες που θα μπορούσαν να ήσαν απάτες. Και το ποσό που αφορούσαν αυτές τις παρατυπίες ήταν 1,5 δις. 72% του ποσού αυτού αφορούσε τις ε, δαπάνες συνοχής. Δηλαδή, ενώ η πολιτική συνοχή είναι περίπου το 1 τρίτο του προϋπολογισμού μας, είναι υπεύθυνη για περίπου τα 3 τέταρτα των ποσών που αφορούν όλες τι περιπτώσεις απάτης. Στον τομέα της συνοχή. οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνε για να έχουν τα ανάλογα και αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τους εντοπισμένου κινδύνους απάτης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν όλη τη διαδικασία διαχείρισης των δαπανών έχοντας ε, πολιτικές κατά της συνοχής, ε, αξιολογώντας τους κινδύνους, ε, συντονίζοντα με άλλες αρχές και να ανταποκρίνονται εάν διαπιστώνουν απάτες, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να στέλνουν και εκθέσεις. Κατά τον έλεγχό μα εστιάσαμε στις διαχειριστικέ αρχές και αξιολογήσαμε εάν έχουν σεβαστεί τις ευθύνες τους καθ' όλη τη διαδικασία της διαχείρισης της ε, προσπάθειες κατά της, των απατών. Και θεωρούμε ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά τον εντοπισμό των κινδύνων και τον σχεδιασμό προληπτικών μέτρων, αλλά πρέπει να κάνουν περισσότερα για την, τον εντοπισμό, την ανταπόκριση και τον συντονισμό. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες. Κατά την διαδικασία εφαρμογής ε, της διαδικασίας αυτής. Τη διαδικασία εφαρμογής της καταπολέμησης των απατών. Πρώτα απ' όλα, βελτίωσαν οι διαχειριστικές αρχές τους κινδύνους απατών κατά την περίοδο 2014-2020, αλλά οι αξιολόγηση τους δεν ήταν πάντα αρκετά τεκμηριωμένες και ορισμένα, πολλά μάλιστα κράτη-μέλη, δεν έχουν καθόλου συγκεκριμένη πολιτική αντιμετώπιση των απατών. Τώρα όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό Έχουμε και καλά και κακά. Οι διαχειριστικέ αρχέ βελτίωσαν τα μέτρα για την πρόληψη, αλλά δεν υπήρξε ουσιώδη πρόοδο, ούτω ώστε να παίζουν ενεργό ρόλο και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίε για τον εντοπισμό των δαπανών. Για παράδειγμα, δεν αξιοποίησαν, αρκετά, δεν αρκετά τα στοιχεία που είχαν, δεν τα ανέλησαν σωστά και δεν υπήρχαν επαρκεί διαδικασίε για να παρακολουθούν και να αξιολογούν την επίπτωση των μέτρων πρόληψη και εντοπισμού. Τέλο, στον τομέα της ε, ανταπόκρισης τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίθηκαν αρκετά σε όλες τις περιπτώσεις που εντόπισαν. Διάφορες διαχειριστικές αρχές <clears throat> δεν ενημερώνουν τα αρμόδια σώματα όταν έχουν υποψίες απατών, για παράδειγμα στην εισαγγελία ή άλλους φορείς δίωξης και δεν συντονίζονται με άλλους φορείς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση των απατών. Επιπλέον, τα διορθωτικά μέτρα συχνά έχουν περιορισμένο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Και οι λειτουργίες των υπηρεσιών συντονισμού της καταπολέμησης απάτης δεν είναι παρκώς καθορισμένες. Επιπλέον, πολλές φορές δεν αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις απατών. Άρα δεν ξέρουμε στην ουσία ποια είναι η ποιότητα των αποτελεσμάτων που αναφέρει η Επιτροπή. Για παράδειγμα, στην έκθεση του 17 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης δεν θεωρούμε ότι αντανακλά πραγματικά το επίπεδο των απατών που πραγματικά εντοπίστηκαν, αλλά μόνο αντανακλούν τις περιπτώσεις που τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να αναφέρουν στην Επιτροπή. Επιτέλους, ε, ε, ε, επιπλέον, κάνουμε μια σειρά από συστάσεις προς τα κράτη-μέλη μέσω της ειδική έκθεσής μας προς τα κράτη-μέλη και την Επιτροπή. Εκεί λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν επίσημες στρατηγικές και πολιτικές για να καταπολεμήσουν τις απάτες, να βελτιώσουν τα μέτρα εντοπισμού χρησιμοποιώντας ε, ανάλυση των δεδομένων που έχουν μέσω των κατάλληλων μεθόδων. Επίσης, η Κομισιόν θα πρέπει να πιέσει τις διαχειριστικές αρχές να αναφέρουν όλες τις περιπτώσει στις αρμόδιες αρχές και να ανθαρρύνουν τα κράτη-μέλη η Κομισιόν πρέπει να ανθαρρύνει τα κράτη-μέλη να διευρύνει τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών συντονισμού κατά των απατών. Στις ε, παραγράφους 81, 88 και 90 της έκθεσής μας καλούμε τους νομοθέτες να λάβουν υπόψη διάφορα θέματα που δεν μπορούμε να θέσουμε στην Κομισιόν λόγω της κατάστασης των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό για τις κοινέ προβλέψεις. Στην παράγραφο 81 τονίζουμε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις και την έγκριση του κανονισμού για τις κοινέ προβλέψεις, οι συνομοθέτες θα μπορούσαν να κάνουν υποχρεωτική την έγκριση των εθνικών στρατηγικών κατά της, ε, των απατών. Στην παράγραφο 88 λέμε ότι η χρήση των σωστών στοιχείων και μεθόδων πληροφορικής θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική, να καταστεί υποχρεωτική. Τέλος, στην παράγραφο 90 τονίζουμε ότι οι συνομοθέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο, όπως άλλους τομείς πολιτικής, να εισαγάγουν συγκεκριμένες κυρώσεις και πρόστιμα για όσους διαπράττουν απάτες κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Όπως για παράδειγμα θα μπορούσαν να μην λαμβάνουν ενωσιακές χρηματοδοτήσεις ή να αποκλείονται από διαγωνισμούς. Θα βοηθούσε πολύ αν τα θέματα αυτά λαμβάνονταν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό των κοινών προβλέψεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Είναι σαφής η εικόνα που μας περιγράψατε πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μαζί μας τον ε, Διευθυντή Φρανκ Σεβέρ. Σας δίνω το λόγο και συνέχεια θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Χριστοφόρου για να σας απευθύνει τα ερωτήματά του. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για, το, αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνέδριου. Ε, we are welcoming very much this report from... Εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή από τη σκοπιά ότι το συνέδριο πραγματικά αναγνωρίζει ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις στο σύστημα ε, ελέγχου και διαχείρισης των δαπανών στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Και θέλω ε, να επισημάνω αυτά που ε, ανέφερε και ο κύριος Γκρέτεν όσον αφορά την, ε, τις περιπτώσεις απάτης ε, στον τομέα της γεωργίας σε σχέση με τις επενδύσεις που έγιναν και τις, τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ξέρετε ότι από το 2014 στο σύστημά μας για τη διαχείριση και τους ελέγχους έχουμε υποχρεωτικό πλέον στοιχείο τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση διαφθορά. Και μάλιστα από το 2014 δώσαμε κατευθυντήριε γραμμέ στα κράτη-μέλη, τους, ε, τους ε, παρήχαμε ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τον προσδιορισμό ε, παραγόντων κινδύνου και για την βελτίωση των εσωτερικών τους συστημάτων ελέγχου. Αυτές οι κατευθύνες γραμμές επίσης συμπεριλάμβαναν και μια σειρά αποζητήματα τα οποία περιλαμβάνει και το συνέδριο στην, στις συστάσεις του, όπως για παράδειγμα ε, η ανάγκη μάλλον τα κράτη, η δυνατότητα των κρατών μελών να μπορούν να θεσπίσουν και πιο αυστηρά μέτρα όσον αφορά την καταπολέμηση διαφοράς και για το σκοπό αυτό μάλιστα παρήχαμε και ένα πρότυπο στα κράτη-μέλη ώστε να μπορούμε να, να προωθήσουμε την υποβολή εκθέσεων σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη και αυτό είναι απαραίτητο για να ε, προωθείται η οριζόντια συστηματική ανάλυση των περιπτώσεων ε, απάτης σε όλους τους τομείς. Και για άλλη μια φορά καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν αυτό το πρότυπο ή ε, για και την ανάκτηση αχρεωστήτως ε, καταβληθέντων ποσών που δρά αποτρεπτικά σε πιθανούς ε, απατεώνες και που βοηθά και τη δουλειά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Και γι' αυτό το σκοπό καλό και όλες τις αρχές και όλες τις φορείς να βρίσκονται σε συνεργασία και μαζί μας και όλα αυτά, όλα αυτά είναι συστάσεις που τις βλέπουμε και στην έκθεση του συνεδρίου και το χαιρετίζουμε αυτό. Επίσης, Κερδίζουμε το γεγονός ότι το συνεδρίο, ότι το συνέδριο <clears throat> αναγνωρίζει ότι η Κομισιόν ε, ε, αξιολογεί και αναλύει τους, ε, τις κινδύνους, αναγνωρίζει τις ε, ε, εκστρατείες ευαισθητοποίησης που έγιναν σε 15, σε 15 κράτη-μέλη για την ανάγκη να υπάρχουν μέτρα κατά της διαφθοράς και της απάτης. Έγιναν και έλεγχοι. Είπα ότι είναι και υποχρεωτική η έλεγχη αυτή. Οι έλεγχοι πλέον από, γίνονται από τα κράτη-μέλη, από την Κομισιόν και αυτοί θα πρέπει πλέον να, ε, ε, ε να αφορούν και το σύστημα ελέγχων. Από πλευράς Κομισιόν κάναμε 22 τέτοιους ελέγχους. Τα κράτη-μέλη όμως είναι υποχρεωμένα να κάνουν ε, Τέτοιου ελέγχου για όλα τα προγράμματα. Επίση, αναθέσαμε εξωτερική μελέτη για ένα δείγμα 15 προγραμμάτων για να δούμε πώς αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται στην πράξη και τι αποτελέσματα φέρνουν. Και τα αποτελέσματα, τα πορίσματα αυτή τη μελέτη που αναφέρονται και από το συνέδριο στην έκθεση ε, ε, είναι πραγματικά συμπληρωματικά προ αυτά που λέει το συνέδριο. Και έχουμε δει ότι αυτό ε, έχει, έχει οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθητοποίηση, ανάλυση κινδύνου, ανταπόκριση και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, ενδιαφέροντα συστήματα ελέγχου ή μηχανισμοί μετριασμού του κινδύνου στα κράτη-μέλη. Ε, στη βάση αυτών των 15 προγραμμάτων που δειγματοληπτικά ελέγχθηκαν και ε, βλέπουμε ότι, ε, ότι στην ε, περίοδο που διανύουμε, 14-20, αυξήθηκε και η αναφορά τέτοιων περιπτώσεων απάντης και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό συνδέεται και με την γενικότερη βελτίωση του πλαισίου. Επίσης, Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τα ενθαρρύνουμε να ενισχύσουν τα συστήματά του. Χαιρετίζουμε τι συστάσει του συνεδρίου, του ελεγκτικού συνεδρίου. Κύριε ε, Γκρέτεν, είπατε ότι ε, κάποιες από αυτές απευθύνονται στην Κομισιόν, κάποιες από αυτές απευθύνονται στα κράτη-μέλη και εμείς βεβαίως τις λαμβάνουμε υπόψη και καλούμε και τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους ε, εκείνες που τα αφορούν. Εφτά συστάσεις αφορούν την Κομισιόν και τον Όλαφ για την ενίσχυση και την προώθηση εθνικών στρατηγικών κατά πολέμης διαφοράς. Επίσης, είμαστε στη διάθεσή σας και στη διάθεση των συνομοθετών για να συνεργαστούμε. Ε, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε κατευθυντήριες γραμμές, βέλτιστες πρακτικές. Ε, σας αναφέρω ενδεικτικά τα εγχειρίδια που έχουμε βγάλει για τα παραποιημένα έγγραφα, για, τις, ε, για τα δύσκολα σημεία σε περιπτώσεις δημόσιων συμβάσεων, τους, τους τομείς κινδύνου και αντίστοιχα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί. Για, το, για την περίοδο μετά το 2020 προβλέπονται απαιτήσει για την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η οδηγία PIF. Όλαφ προωθεί και έναν ευρύτερο λόγο τον, ε, ρόλο των ΑΦΚΟΣ και η τελευταία σύσταση στην οποία συμμετέχουμε, ε, συμφωνούμε εν μέρη μόνο την ανάγκη αξιολόγησης των μέτρων ε, κατά ε, καταπολέμησης διαφθοράς και της απάτης. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ε, ευρύ και πάρα πολύ περίπλοκο ως ε, καθήκον. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σύσταση για το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ο Όλαφ, ωστόσο, έχει αναθεωρήσει και επικαιροποιήσει τη στρατηγική της Κομισιόν για την καταπολέμηση της διαφθοράς και καταρτίζει και προφίλ κατά κράτος σχετικά με τις ικανότητες που χρειάζονται και που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν στην περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ κύριε Γκρέτεν, κύριε Ισηγητά και κύριε Πρόεδρε για τον λόγο. like to the Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Χριστοφόρ και στη συνέχεια στη σκιώδη Ισηγήτρια, την κυρία Κινίτση. Σε λίγα λεπτά θα, θα τελειώσει και η διερμηνία, οπότε να δώσω τον λόγο στους δύο συναδέλφους να μιλήσω στη γλώσσα τους. Ο κύριος Χριστοφούρ φόρου, λοιπόν παρακαλώ όσο γίνεται πιο σύντομα να μας τα πει. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Πρόεδρε, να... θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω και τον αγαπητόν Χέριν Κρέντεν και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ιδιαίτερα σημαντικές επισημάσεις και διαπιστώσεις. Εγώ μπορώ να πω σε όσα υπόθηκαν δεν έχω να προσθέσω οτιδήποτε. Είναι διαπιστώσει και επισημάσει που όλοι συμφωνούμε και είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η έκθεση που ουσιαστικά επικεντρώνεται εκεί που πραγματικά έχει πρόβλημα ο έλεγχος και έχει πρόβλημα στην κατασπατάληση ε, ευρωπαϊκού χρήματο που είναι οι πολιτικέ συνοχή. Φυσικά, αν κάποιο δει στο, στο ποσό του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ που είναι το 75 που αφορά τη συνοχή ως ποσοστό επί του συνόλου των προπολογισμών είναι πολύ μικρό. Όμως έστω και έναν ευρώ να χάνεται σε ζητήματα απάτης εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Είμαι ιδιαίτερα όμως απεσιόδοξο σε ένα σημαντικό σημείο. Η έκθεση προβαίνει σε επισημάσεις ότι οι εθνικές διαχειριστικές αρχές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο να εφαρμόσουν εθνική στρατηγική the translation or the asking to slow down a little bit Όμως μέσα στην έκθεση την ιδιαίτερα σημαντική και επικροτώ ξανά όσα αναφέρονται υπάρχουν διαπιστώσεις. Το θέμα είναι πώς υλοποιούνται αυτές οι διαπιστώσεις για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή όταν αναφέρεται ότι οι εθνικές διαχειριστικές αρχές καταπολέμησης της απάτης είναι ανεπαρκείς, δεν ανταποκρίνονται τα κράτη δεν επιδεικνύουν τον ε, αναμενόμενο, το αναμενόμενο ενδιαφέρον για να προβούν στην καταπολέμηση της απάτης. Εμείς πώς ανταποκρινόμαστε ούτως ώστε να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη και γιατί πρέπει το κάθε κράτο μέλος να υποχρώνεται από μόνο του να εφαρμόσει αυτή την αρχή και να μην υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχή καταπολέμησης της απάτης που θα θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι κοινοτικό και χτυμένο και θα απεχρώνονται τα κράτη-μέλη να το εφαρμόσουν. Θα μπορούσε να μπει μια γενική αρχή ότι δεν παραχωρείται ούτε έναν ευρώ σε καμία χώρα μέλο εάν δεν εφαρμόσει αυτή την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση τη απάτη. Να φύγουμε από την αρχή ότι δίνουμε χρήματα και περιμένουμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα. Πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του να προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα και προ αυτήν την κατεύθυνση πρέπει ουσιαστικά ε, να κινηθούμε όλοι μα. Θέλω να ρωτήσω όμω, ένα βασικό ζήτημα είναι τα μέτρα πρόληψη τη απάτη. Ένα μέτρο πρόληψη τη απάτη είναι αυτή η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική και γιατί δεν εφαρμόζεται. Σίγουρα δεν ευθυνεται ούτε το ελεκτικό συνέδριο και πιθανώ ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπάρξει κοινή προσπάθεια. Δεύτερο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι απάτε πρέπει να έχουν κόστος αποτροπής. Και ένα βασικό κόστος αποτροπής είναι το πολλαπλάσιο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλεται. Γιατί δεν υποχρώνουμε να επιβάλλονται αυτά τα πρόστιμα. Τρίτο και σημαντικό είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών μέσων που σήμερα σε μια ψηφιακή εποχή θα μπορούσαμε να προλαβαίνουμε αυτές τις απάτες. Ταυτόχρονα θα ήθελα να γνωρίζω αν οι ελεκτικές αρχές, ο Όλαφ, έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή του είναι επαρκή σε ανθρώπινο δυναμικό, σε προπολογισμό, σε τεχνικά μέσα, σε ψηφιακά μέσα για να μπορέσει να προλαβαίνει αυτέ τι απάτε και να αποτελεί πραγματικά στοιχείο αποτροπή. Σημασία δεν έχει να τρέξει να αποκαταστήσει μια απάτη που έγινε που όπω αναφέρει η έκθεση χρειάζεται πολλή χρόνο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί μια απάτη και στο τέλο, να τιμωρηθεί αυτό που τη διέπραξε που αυτό αποτελεί κίνητρο για του απαταιώνε εμείς με ποιον τρόπο μπορούμε να αποτρέψουμε και να μειώσουμε και να περιορίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν μια πολύ σημαντική έκθεση. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση είναι καθοδηγητή μα, όμω πιστεύω πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα προ τι χώρε μέλη, ούτω ώστε στην επόμενη έκθεση να μην χρειάζεται να μιλάμε για 1,5 δισεκατομμύριο ε, κόστο τη απάτη. Ευχαριστώ. Vielen herzlichen Dank. Ich darf nun Katharina Kinitschi das Wort geben. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Γκρέντενα. Ε, ευχαριστούμε τους φιλοξενουμένους μας για τα όσα μας παρουσίαν. Πολύ σημαντικό το θέμα για τις χώρες. Και νομίζω ότι η σύνοχη πραγματικά είναι πολύ ε, σημαντική για όλους. Άρα θα πρέπει να σταματήσουμε τις απάτες σε σχέση με τους πόρους της συνοχής. Είναι απαραίτητο και επίσης απαραίτητο να κάνουμε διόρθωση πορείας και να μην συμβαίνουν τέτοιες απάτες. Ήδη το είπαμε και το ξαναείπαμε ε, για περιοριστώ λοιπόν σε κάποιες ε, σκέψεις. Πρώτα πρώτα ξέρουμε ότι ε, εν μέσω των κρατών μελών δεν υπάρχει κοινό ορισμός. Αυτό είναι ανομαλία. Άρα θέλω αυτό να το διορθώσουμε, να υπάρχει ενιαία ερμηνεία, ενιαίος ορισμός, γιατί αλλιώς είναι ε, φραγμός στο να εφαρμοστεί το κοινωτικό δίκαιο σε αυτόν τον τομέα. Άρα θα πρέπει να το τσεκάρουμε το θέμα. Επίσης γνωρίζουμε ότι σε κάποια κράτη-μέλη δεν έχει υιοθετηθεί επίσημη πολιτική κατά της απάτης. Άρα και εδώ θα πρέπει, ε, όπως είπε ο συνάδελφος, να λάβουμε υπόψη το, την αρχή της επικορικότητας για να δούμε τι μέτρα μπορούν να θεσπίσουν τα κράτη-μέλη για μια τέτοια πολιτική, επίσημη πολιτική κατά της απάτης. Να δοθούν όλα τα στοιχεία στην Επιτροπή, γιατί δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό από όλες τις χώρες. Και ξέρουμε ότι πολλές χώρες δεν χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης αυτών των δεδομένων. Έχουμε και το σύστημα ράκνε. Εργαλείο που θα πρέπει να επισημοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Κομισιόν και έτσι θα έχουμε το κίνητρο χρήσης του μηχανισμού. Τελευταίο θέμα. Γρήγορα, γρήγορα, Τελευταία Τελευταίο, τελευταίο. Ερώτηση συγκεκριμένη. Αναδείτε στην έκθεση το πώς οι διαχειριστικές αρχές έχουν κάποιες μεθόδους άτυπες για να επισημάνουν τις απάντες σε χώρες. Και υπάρχουν δυσκολίες δυσκολίες, πολλές φορές είναι και θέμα νοοτροπίας. Το, θέμα των καταδοτών, των whistleblowers. Όμως αυτό βοηθά σημαντικά. όλα έχουμε την οδηγία, το πριν το 19, έτσι, έχουμε μείζονες εγγύησεις όσον αφορά την προστασία αυτών των μαρτύρων, αυτών των πληροφοριδοτών. Τι λέει το συνέδριο αρκούν αυτά τα μέτρα. Τι λέει η Κομισιόν. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στις χώρες. Να χρησιμοποιήσουν καλύτερα αυτά τα μέσα, τα εργαλεία. Πώς θα οθήσουμε τα κρατημέλεια να υιοθετήσουν το νωρίτερο δυνατόν την οδηγία. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich darf vielleicht noch kurz Katharina Gschee bitten, muss allerdings sagen, dass jetzt die Übersetzung aufhört, aber sie spricht perfekt Englisch, soweit ich das weiß